Καλημέρα σας. Ladies and gentlemen, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε. Αργήσαμε ήδη 10 λεπτά. Περίμενα τα μέλη της Επιτροπής. Ο εισηγητής είναι εδώ, οπότε μπορούμε και να αρχίσουμε. Παύλο Σάλβα. Και ο κύριος Λάγκη είναι εδώ. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το σημείο 15 της μερισίας διάταξης. Διμερείς ε, ρήτρα διασφάλισης ε, και μηχανισμού σταθεροποίηση για τι μπανάνε στο πλαίσιο τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κολομβία και Περού. Και στη συνέχεια θα περάσω. Ε, ο εισηγητή, συγγνώμη, είναι ο κύριο Μπέρντ Λάγκε. Έχετε στου φακέλου σα το σχέδιο της πρότασης και τη μελέτη σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες. Ε, Μπεν, θα σου δώσω το λόγο για να εισαγάγεις το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών, όπως και στην περίπτωση της ε, Νότιας ε, Κορέας, υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ρήτρα ασφαλείας, ο οποίος, αγαπητοί συνάδελφοι, μοιάζει πάρα πολύ με το μηχανισμό που προβλέπεται στη Συμφωνία με τη Νότια Κορέα. Έτσι λοιπόν στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση οποτεδήποτε πρόκειται για απρόβλεπτες ε, καταστάσεις, ε, γεγονότα μπορεί να πυροδοτηθεί ένας ε, μηχανισμός για να προστατευτούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Δηλαδή προβλέπεται η δυνατότητα να επανέρχεται η επιβολή δασμών. Όπως ε, σας είπα, ο μηχανισμός αυτός ε, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που χρησιμοποιείται για την Νότια Κορέα. Βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα που είναι ξεχωριστό, αφορά τις μπανάνες. Εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε μια ειδική ρύθμιση η οποία προβλέπει σύστημα ποσοστώσεων έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μπανάνας να προστατεύονται ιδιαίτερα και να έχουν τη δυνατότητα τους παραγωγούς από απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να τους προστατεύουν ιδιαίτερα. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία οφείλουμε να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας. Ε, συνολικά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, τίθεται το εξής ερώτημα. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι εφαρμόσιμο και πότε εφαρμόζεται. Αυτό ε, συνδέεται αφενός με το ότι η γραφειοκρατία και οι δαπάνε είναι αρκετά υψηλέ. Γι' αυτό λοιπόν αυτό ο μηχανισμό σπάνια εφαρμόζεται. Και δεύτερον, μοιάζει με άλλου μηχανισμού που έτσι κι αλλιώ προβλέπονται. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι πολύ συχνά δεν γίνεται χρήση αυτού του μηχανισμού. Και εκτό αυτού πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε το ε, πώς ακριβώς μπορούμε να καταστήσουμε πιο εύκολο εφαρμόσιμο αυτό το εργαλείο. Ε, καταρχήν, τίτε το ερώτημα πότε ισχύουν αυτοί οι κανονισμοί ασφαλείας. Ποιο είναι το κριτήριο. Και εδώ ισχύει το εξής. Αυτό το, αυτός ο μηχανισμός επηρεάζει ιδιαίτερα, μάλλον ισχύει ο μηχανισμός όταν ε, ασκούνται μεγάλες ε, επιρροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δούμε την Κολομβία, παραδείγματο χάρη, τότε τίθεται το ερώτημα κατά πόσον πράγματι εδώ πρόκειται για ε, το σωστό εργαλείο. Γιατί ε, αν δούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσον μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα άλλο μέσο. Δεύτερον, ποιος μπορεί να εισάγει έρευνα. Αυτό το συζητήσαμε επανειλημμένα σε σχέση με τους ε, κανονισμούς ε, ρήτρας ασφαλείας ε, που ισχύουν για την Νότια Κορέα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ισχύει και εδώ το ίδιο, όπω ισχύει και με την Νότια Κορέα. Να παρακολουθούμε δηλαδή τι εξελίξει ε, στο κράτο και η Κομισιόν να προβαίνει σε μια ιδιαίτερη δήλωση. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε το κατά πόσον ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, τόσο δηλαδή με τους παραγωγούς ε, όσο και με εκείνους που εργάζονται στο τομέα, κατά πόσον ο διάλογος αυτός μπορεί να ενισχυθεί. Και Βεβαίως ε, τίθεται και το ερώτημα του τομέα της ε, μπανάνας. Για μένα δεν είναι απόλυτα σαφές το πιο ακριβώς ε, πρέπει να είναι το κριτήριο για, τον, για την ποσότητα και επίσης και ποιο έτος λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς υπολογισμού ποσοστώσεων για τις μπανάνες. Πρέπει επίσης να δούμε ποια είναι η ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στη ρήτρα ασφαλείας για τις μπανάνες και ε, γενικότερα την διατύπωση ρητρών ασφαλείας. Πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, η σχέση ή αυτά που ορίζουμε είναι εφαρμόσιμα ή μήπως θα πρέπει να προβούμε σε μια ιεράρχηση. από τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που παράγουν μπανάνες άκουσα αρκετή κριτική και ισχυρίζονται οι χώρες παραγωγή ότι αυτά τα οποία προβλέπονται δεν είναι εφαρμόσιμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ε, ερωτήσεις ε, και μερικοί μας παροτρύνουν να βελτιώσουμε την ισχύουσα πρόταση. Πολλοί ρωτάνε τελικά υπάρχει κάποια εμπειρία με αυτή τη ρήτρα ασφαλεία ε, με τη Νότια Κορέα. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να τοποθετηθεί από αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εφαρμογή της ε, ρήτρα ε, διασφάλισης στη συμφωνία με την Κορέα. Πριν να αρχίσουμε την συζήτηση, Θα ακούσουμε το σκιώδη από την Επιτροπή Γεωργίας για αυτό το θέμα. Γκαμπριέλ Μάτσα, έχουν ε, εκδώσει γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γεωργίας. Είστε εδώ κύριε Μάτσα, παρακαλώ μπορείτε να μας ε, την παρουσιάσετε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ και μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ε, θέση μας εδώ στην Επιτροπή σας ΙΝΤΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα τον κύριο Λάγκε για την ε, παρουσίασή του. Τώρα να σας πω ευθύ εξ αρχής ότι από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας είναι προφανές ότι έχει συναπόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ε, ενσωμάτωση της νομοθεσίας. Όμως δυστυχώς είναι μάλλον εικονική η εξουσία αυτή γιατί οι ρήτρε αποτελούν μέρος των συμφωνιών και στη διαπραγμάτευση αυτών απουσιάζει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε να συμμετέχει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις που γίνονται με τρίτες χώρες γιατί αυτές οι, συμφωνίε οι συμφωνίες νόμοι έχουν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, κάτι το οποίο πιστεύω αιτιολογεί απόλυτα να παίζει πιο ενεργό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εσείς, η Επιτροπή σας, θα μπορούσε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο αίτημα αυτό, προκειμένου να συμμετέχει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται εν ώψη των εμπορικών αυτών συμφωνιών. Τώρα το Κοινοβούλιο παρεμβαίνει υπερβολικά αργά και οι ρήτρε ε, ασφαλείας είναι τέτοιες που δεν βοηθούν παρά μόνο στο θέμα της μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Το περιθώριο λοιπόν ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ περιορισμένο. Πιστεύω όμως παρόλα αυτά ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ε, τα όσα θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς όμως να τροποποιήσουμε και το πνεύμα των συμφωνιών με τρίτες χώρες. Αυτό ε, πιστεύω ότι προσπαθεί να κάνει και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας. Τι προτείνω εγώ λοιπόν. Πρώτον, να αφαιρεθούν, ε, μάλλον να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις οποιοδήποτε στρεβλώσεις μπορεί να δημιουργούνται στην αγορά. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω κάτι που πιστεύω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμφωνία με την Κολοβία και το Περού. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην ε, Νότια Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι που μας ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερως εδώ. Οι συμφωνίες αυτές έχουν τεράστιες επιπτώσεις στα γεωργικά προϊόντα θέλουμε μεγαλύτερο άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε προϊόντα όπως είναι η μπανάνα, το βόλιο κρέας και η ζάχαρη. Ενώ, το Ευρω... ενώ η Ευρώπη από τη δικιά της την πλευρά μπορεί να βοηθήσει με το γάλα, τα δημητριακά και το χείριο κρέας που εξάγει προς τις χώρες αυτές. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο αναγνώρισης των ονομασιών ποιότητας. Αυτό είναι πολύ θετικό πιστεύω. Τώρα η μπανάνα βλέπετε ότι αποτελεί και ε, το, τη στάρα ας πούμε, της διαπραγμάτευσης αυτής. Ο περιορισμός των δασμών που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εισαγωγές από πλευράς των Ευρωπαίων παραγωγών ε, φαίνεται ότι πλήττει τα δικά τους τα συμφέροντα. Γι' αυτό και προβλέπεται ένας μηχανισμός με στόχο να αποφευθεί η εισαγωγή φρούτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπερνάνε κάποιο όριο. Ο μηχανισμός θα βοηθήσει ε, να μην υπάρχουν οι δασμοί ανάλογα με τις ποσότητες, αλλά αυτό μόνο για μια ανώτατη περίοδο τριών μηνών. Επιπλέον, ο μηχανισμός αυτός προβλέπει και κάτι σημαντικό. Ο κύριος Λάγια αναφέρθηκε σε αυτό, χωρίς να καταλαβαίνει πολύ καλά. Ε, λοιπόν, τα ποσοστά που προβλέπονται στη ρήτρα έχουν υπολογιστεί προς τα πάνω. Είναι δύσκολο η αγορά να πλήττεται από στρεβλώσεις ακόμα και πριν να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Πάντως αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί για την Κολοβία και την Κωνσταντίνα που είναι οι δύο χώρες με περισσότερες εξαγωγές, βλέπετε διπλασιάζονται οι ποσοστώσεις. Δεν ξέρω σε τι όγκο ακριβώς, πάντως αυτό το οποίο προβλέπετε είναι να διπλασιαστεί η ποσότητα, κάποια εκατομμύρια τόνοι. Οι στρεβλώσεις δηλαδή μπορεί να προκληθούν πολύ πριν καταλήξουμε στη συμφωνία. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε. Η θέση σε ισχύ του μηχανισμού δεν είναι αυτόματη. Δηλαδή η Κομισιόν τι λέει. Λέει ότι μπορεί να μην θέσει σε ισχύ τον μηχανισμό εφόσον ε, διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες ε, προκαλούν ζημία κλπ. Εγώ το πρόβλημα πάντως που βλέπω ξεκάθαρα είναι ότι το σχέδιο μηχανισμού μπορεί να οδηγήσει σε ένα περιθώριο διακρίσεων το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και το οποίο πρέπει να περιορίσουμε έτσι ώστε να προστατεύσουμε όσο γίνεται καλύτερα την ευρωπαϊκή παραγωγή. Λοιπόν, να μην είναι στη διακριτική ευχέρεια ε, κανενός. Αναφέρομαι τώρα στο άρθρο 13. Πιστεύω ότι μόνο σε περίπτωση ε, ύψης ανάγκης πρέπει να μνήσει ο μηχανισμός. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τίθεται σε ισχύ ο μηχανισμός αυτός. Κάτι άλλο είναι η ενίσχυση του μηχανισμού σταθεροποίησης προκειμένου να χρησιμεύσει σαν ε, καμπανάκι κινδύνου για να υιοθετούνται τα κατάλληλα μέτρα διόρθωσης. Όπως προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής, ο μηχανισμός σταθεροποίησης της Βανάνας είναι από δίπλα, δεν συνδέεται με τίποτα με τη ρήτρα ε, διασφάλισης. Εμείς και εγώ θα ήθελα η έκθεσή μας να κάνει ακριβώς το αντίθετο, να συνδέονται οι δύο μηχανισμοί. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ βασικό. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, στο άρθρο 4 του κανονισμού, εκεί που λέμε ότι μόλις ε, φτάσουμε στο ποσοστό του μηχανισμού πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες και τη ρήτρα διασφάλισης. Τι θέλουμε με αυτό, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ρήτρα θα εφαρμόζεται εφόσον χρειαστεί και στο τομέα της μπανάνας. Πρόκειται δηλαδή για κάτι το οποίο ξεπερνά το μηχανισμό σταθεροποίησης και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα στην ρίζα του. Όπως είπα και πριν, εάν ο μηχανισμός ισχύει τρεις μήνες, η ρήτρα μπορεί να ισχύσει δύο ε, χρόνια και μάλιστα να παραταθεί επίσης. Στο άρθρο 13 τώρα μιλάμε για μέτρα πρόληψης που περιλαμβάνονται στη ρήτρα διασφάλισης εφόσον έχει επιτευθεί ο όγκος ε, ο οποίος θέτει σε ισχύ το μηχανισμό. Θα ολοκληρώσω με το εξή. Η εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίησης δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα ούτε πρέπει να δυσκολεύει την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στη ρήτρα διμερούς διασφάλισης για τον τομέα της μπανάνας. Η έκθεση πάντως που παρουσιάζεται στην Επιτροπή πρέπει να υπογραμμίζει και τη σημασία που έχει το να παρακολουθούμε τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Μπανάνας για να αποφεύγουμε στρεβλώσεις στην αγορά και να μπορούν να εφαρμόζονται οι διατάξει διασφάλισης έτσι όπως έχουν προβλεφθεί όταν καλύπτονται οι προϋποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να παρακολουθούμε τις εξαγωγές που κάνουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και άρα η Κομισιόν πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες με τα κράτη-μέλη αφενός, από την άλλη μεριά όμως και με την, τον αντίστοιχο κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα τι κατάσταση επικρατεί στην αγορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα και με ίδια πρωτοβουλία θα πρέπει να ε, εφαρμόζει ε, έγκαιρα τα μέτρα που προβλέπονται στην ρήτρα. Τέλος υπάρχει και μια παρουσίαση για ετήσια ε, παρουσίαση της κατάστασης όσον αφορά την μπανάνα και της ευρωπαϊκής παραγωγής μπανάνας. Θα έπρεπε πληροφορίες να είναι λεπτομερείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορούμε να τις έχουμε κάθε φορά που τις ζητάμε βάσει των στοιχείων που ακριβώς έχουν συμπεριληφθεί στην ετήσια έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Μας αρχίσουμε τη συζήτηση. Χωσέ Ανδρέα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Λάγκε για τα όσα μας είπε. Στη συμφωνία αυτή αναφέρεται η αμοιβαιότητα. Υπάρχει η ρήτρα διασφάλισης, όπως έχουμε και με την ε, Κορέα και με το Μαρόκο. Τι προσπαθεί να πετύχει η ρήτρα αυτή διασφάλισης. Θέλει να δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό που να αποφεύγει την αποσταθεροποίηση στην αγορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως τώρα της μπανάνας, έχει να κάνει με ιδιαίτερα περιφερειακές και ευαίσθητες περιοχές που εξαρτώνται από τη μονοκαλλιέργεια της μπανάνας, όπου όλο το εργατικό δυναμικό δηλαδή απασχολείται στον κλάδο αυτό και έτσι πολύ γρήγορα κινδυνεύει να υπάρξει αποσταθεροποίηση. Γι' αυτό και πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε, όπως έλεγε ο κ. Μπάρτο, πολύ γρήγορα βάσει μιας ρήτρα διασφάλισης η οποία να ελέγχει πρώτα, βάσει της οποίας να ελέγχεται πρώτα η κατάσταση και αμέσως μετά να μπορεί να υπάρξει δράση για σταθεροποίηση στην αγορά. Υπάρχουν και προηγούμενα όπου κάθε μήνα γινόταν σχεδιασμός των ποσοτήτων που εισάγονταν, όπως για παράδειγμα με το Μαρόκο. Οπότε και εδώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει το ίδιο σχεδιασμό δηλαδή των ε, ποσοτήτων ε, μπανάνας που μπορούν να εισαχθούν για να ξέρουμε πώς θα επηρεαστούν οι άκρος περιφερειακές περιοχές οι οποίες ζουν από την μονοκαλλιέργεια αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα έπρεπε να είχα αρχίσει από έναν άλλο μιλητή. Δεν θέλετε το λόγο. Ναι, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τόσα είπαν ε, οι συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κάθριν δεν είναι εδώ. Ε, ε, από την παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγήτη και τον Σκιώδη από την Επιτροπή Γεωργίας διότι όντω αυτά τα θέματα ρητρών διασφάλιση ε, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Ε, πραγματευόμαστε αυτά τα πολυσύνδετα ζητήματα της ρήτρας ε, διασφάλισης ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα ζητήματα με τη Γενική Συμφωνία. Ε, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τη δινή οικονομική κατάσταση των χωρών για τις οποίες ε, συζητάμε, αλλά και την ε, οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ακολουθούμε τη γραμμή του εισηγητή εν γέννη και θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το επιχείρημα που μόλις ανέφερε ε, η Νομισματική Επιτροπή σημείωσε επιτυχές εργασίες της, ε, η Επιτροπή δηλαδή που ε, συγκροτήσαμε. Υπάρχει μία ε, συνένεση, αν θέλετε, για τα ζητήματα. Και η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ώστε να βρεθεί μια συμβαστική λύση με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τη Γραμματεία για την υποστήριξη Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ρόμπερτ Στέρντι, Ρόμπερτ Στέρντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι την πολυπλοκότητα του ζητήματος και ευχαριστώ τον εισηγητή για ό,τι έκανε. Η πραγματική μου ανησυχία έγκυται στο εξή. Η Επιτροπή, με Επιτροπή Εμπορίου δεν μπορεί να ε, εμπλακεί σε απόπειρε προστατευτισμού. Θέλω λοιπόν να αποφύγουμε αυτήν την κατάσταση συγκρότηση ενό μηχανισμού που έχει σχεδιαστεί ε, για δασμολογικού φραγμού ε, ή για σκοπού προστατευτισμού. Εγώ επί σειρά ετών ασχολήθηκα με τι συμφωνίε για τη ζάχαρη ε, και έλεγαν όλοι όλα εκτός από την ε, μπανάνα και εκτός από την ε, ζάχαρη. Και τα ίδια προβλήματα είχαμε και με τις χώρες ΑΚΕ γιατί ήμουν μέλος της Επιτροπής και παρακολούθησα εκ του σύνεκης τον παραγωγικό μηχανισμό για τις μπανάνες και τελικά συνήθι μια κακή συμφωνία. Αυτό που με ανησυχεί εδώ είναι ότι ο μηχανισμός αυτός ταυτίζεται με πλήρη προστατευτισμό για ολόκληρο κλάδο της αγοράς. Είμαι σίγουρος δεν θα με υποστηρίξετε, αλλά θα το πω. Θα πρέπει να εξετάσουμε ανταυτού το εξή. Μήπω μπορούμε να συγκροτήσουμε έναν ε, ε, μηχανισμό κοινωνικού χαρακτήρα για αυτού του ανθρώπου, να του προστατεύσουμε ένα σύστημα που όχι απαραίτητα του προστατεύει, αλλά του επιτρέπει να ανταγωνίζονται πιο ελεύθερα στι ε, διεθνεί αγορέ. Στην κοινή γεωρική πολιτική θέλουμε να απομακρυνθούμε από τα επιδόματα, από το, του μηχανισμού στήριξη. Πλην όμω, υπάρχουν κάποιε χώρε όπου ίσω χρειάζονται ακόμη επιδοτήσει, ούτω ώστε ε, να, ανθεί, να συνεχίζει να ανθεί ε, η γεωργία. Ε, φοβούμε λοιπόν γιατί είναι υπερβολικά προστατευτικό σε εισαγωγικά το κείμενο. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Στέρντι. Ποιο άλλο θα ήθελε το λόγο. α ακούσουμε τότε τον τον Τζον Κλάρκ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πού είστε και ποιος είστε. Ε, πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Και εγώ αναρωτιέμαι το πρωί ποιο είμαι. Είμαι επικεφαλή ε, ε, του ε, τμήματο άμυνα εμπειρική πολιτική στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Trade. πολύ πλούσια συζήτηση και πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα και τα επιχειρήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Όντω αληθεύει ότι αυτή η αναχείρα πρόταση απορρέει σε μεγάλο βαθμό από τον κανονισμό, το βασικό κανονισμό για τι ρήτρε διασφάλιση που έχουμε συζητήσει εκτενώ και σε τριμερεί διαλόγους και στην Επιτροπή το 2010 κυρίως. Ως εκ τούτου διαθέτουμε μια, ένα πάρα πολύ καλό έρισμα για την εκπόνηση της νέας πρότασης που τώρα εξετάζει η Επιτροπή. Θα άξιζε ίσως να υπενθυμίσουμε ποιος είναι ο στόχος αυτών των μηχανισμών διασφάλισης. Ο στόχος τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ε, βάσει τη απελευθέρωση του εμπορίου και αύξηση ε, των εισαγωγών που πλήττει τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούμε να επιστρέψουμε στην ρήτρα για το Most Favored Nation, το πλέον ευνοούμενο κράτος Υπάρχουν όργανα, εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να ρυθμίσουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το dumping, παραδείγματος χάρη, ή την κατάργηση των επιδοτήσεων που χρησιμοποιούνται από τα θεσμικά όργανα σε τακτική πλέον βάση. Κάποια μέλη της Επιτροπής ανησυχούν ότι τα εργαλεία αυτά που θα χρησιμοποιηθούν ε, ίσως κρύβουν εκπλήξεις γιατί δεν έχουν ξεχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν αληθεύει ότι στο, μέτρο, στο παρελθόν δεν είχαμε αντίστοιχη ρήτρα διασφάλισης. Μάλλον προβλεπόταν στην κείμενη νομοθεσία, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Η βιομηχανία ε, έχει ζητήσει την εφαρμογή αυτής της ρήτρα. Για τον εξής λόγο, η ευρωπαϊκή δασμή είναι σχετικά χαμηλή και άρα περαιτέρω μείωση ή άρση των φραγμών ουσιαστικά δεν δημιουργεί προβλήματα στη βιομηχανία διότι η βιομηχανία έχει ήδη συνηθίσει, είναι εξοικειωμένη δηλαδή με τον διεθνή ανταγωνισμό. Τούτου λεχθέντος ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία και έχουν σχεδιαστεί επί τη βάση ενιών και διαδικασιών που υπακούν στην επιταγή της καταπολέμησης του ντάμπινγκ. Αλλά όπως είπα, χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια αυτά τα εργαλεία. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατακαιρματισμένες βιομηχανίες, διότι μπορεί να ε, επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες τεχνικές. Δημιουργείται λοιπόν μια ζώνη ασφαλείας. Αυτή η ζώνη ασφαλείας όπως και στο αυτοκίνητο ε, ε, είναι χρήσιμη όταν υπάρχει ένα ατύχημα. Ε, ο στόχος ήταν να υπάρχει ένας μηχανισμός διασφάλισης για καταστάσεις επίγουσας ανάγκης. Κάναμε και τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών. Προτού συντάξουμε την πρότασή μας Ε, αλλά ε, ξαναλέω ότι είναι περιορισμένου εύρους οι ρήτρες διασφάλισης ε, και τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα κοινωνικά ζητήματα τα πραγματευόμαστε σε διαφορετικό τμήμα του κανονισμού για τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους. Ως προς τα εργασιακά δικαιώματα φροντίζουμε ούτω ή άλλω, διότι υπάρχει η καθολική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλύπτει αυτά τα δικαιώματα και ούτως ή άλλως βάσει τις ρήτρες του Most Favored Nation, του πλέον ευνοούμενου κράτους ε, μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Υπάρχουν ε, διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις, διεθνώς αναγνωρισμένα εργατικά δικαιώματα και προβλέπεται και μηχανισμός διαμεσολάβησης. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί και αυτά είναι τα φόρα, τα βήματα που θα πρέπει να καλύψουμε μέσα στην πρόταση, να μην περιοριστούμε δηλαδή σε, αυτά τα, σε αυτές τις διμερείς ε, ρήτρες διασφάλισης ε, που αποσκοπούν, το ξαναλέω, ε, στη ρύθμιση εκτάκτων περιστώσεων. Κάτι άλλο τώρα. Ποια η σχέση ανάμεσα στον μηχανισμό, το διμερή μηχανισμό ρήτρες διασφάλισης για την μπανάνα και την γενικότερη διμερή ρήτρα διασφάλισης, όχι για την μπανάνα, που υπάρχει σε όλα τα νομικά εργαλεία. Ο μηχανισμός για την μπανάνα είναι το πλέον πρόσφορο εργαλείο. Όμως αυτό δεν αποκλείει άλλες περιπτώσεις χρήσης του διμερούς μηχανισμού διασφάλισης το πνεύμα που διαπνέει αυτά τα εργαλεία, η εφαρμοστική όρη καθώς και η διάρκεια των μέτρων από οποιαδήποτε από αυτά τα εργαλεία ε, διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό. Αν θέλετε να δημιουργήσετε τον διμερή μηχανισμό πρέπει να αποδείξουμε ότι λόγω της απελευθέρωσης των δασμών και της αύξησης των ε, εισαγωγών έχει πληγεί η βιομηχανία. Πρέπει φυσικά να γίνει έρευνα που διαρκεί έξι μήνε πρωτού στοιχείο. Και φυσικά για δύο χρόνια μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα και δυνατότητα διετού ανανέωση. Η διαδικασία αυτή είναι θελκτική, ας το πω έτσι. και έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις επί του εμπορίου. Σχετικά τώρα με τη ρήτρα διασφάλισης της μπανάνας. Πολύ απλούστερος αυτός ο μηχανισμός. Ποιο είναι το εφαλτήριο. Αν φτάσουμε έναν όγκο ενεργοποίησης του μηχανισμού και μετά από διαβούλευση με τις χώρες εταίρους και εξετάζοντας τις ιονή αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμεθα για μια σχετικά βραχία περίοδο να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον μηχανισμό και επιστρέφουμε στο δασμό MFN για τρει μήνες. Επίσης, ε, μα ζητήθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να προσδιορίζουμε και τον όγκο ενεργοποίηση του μηχανισμού, τον όγκο εμπορευμάτων που ενεργοποιεί τον μηχανισμό. Ε, αυτά ως προς την εφαρμογή. Παρατηρείτε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στους δύο. Θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης ε, τις επιπτώσεις κατά περίπτωση όταν ε, αποφασίζουμε ενεργοποίηση ε, ε, κάποιου μηχανισμού. Τώρα, ας περάσω στο θέμα της Κορέας. Ως προς την εφαρμογή της, του διμερούς μηχανισμού διασφάλισης, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στο παρελθόν με την Κορέα. Παρακολουθούσαμε τα ιδιαίτερα ευάλωτα προϊόντα. Έχετε λάβει ε, τη σχετική έκθεση αξιολόγηση, ε, ενημερώνεται και η βιομηχανία. Μέχρι τούδε δεν έχει σημειωθεί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν ζήτησε ενεργοποίηση του μηχανισμού διασφάλισης βιομηχανία. Σταματάω εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τον εισηγητή μας, ε, Μπέντ Λάγκη, για τις τελικές παρατηρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους ε, συναδέλφου ε, για τις προτάσεις τους. Νομίζω ότι κατέστη απόλυτα σαφέ, ότι όσον αφορά το θέμα των ποσοστώσεων και των κριτηρίων για την έναρξη ερευνών, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε πράγματι να αποκτήσουμε σαφήνεια και αυτό ισχύει κυρίως ε, για την μπανάνα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δυναμικό βελτίωσης ε, έτσι ώστε να μην πρόκειται απλά και μόνο για ε, ζώνες ασφαλείας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μερικές φορές δεν τις φοράει κανείς τις ζώνες ασφαλείας και είναι και άχρηστες. Δεν θέλω να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο το εργαλείο μας. Αναφέρομαι τόσο στο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να το ξανασκεφτούμε, όπως ε, και ε, στα κριτήρια. Και επίσης, ε, κύριε Μιούλα, δεν νομίζω ότι πρέπει να μας επισημαίνετε ότι στο θέμα αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ευρωβουλευτές. Εκείνο το οποίο τίθεται ως ερώτημα είναι ε, κατά πόσον η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη μπορεί να εκφραστεί περισσότερο και να ακουστεί η άποψή τη για το κατά πόσον θα πρέπει να ξεκινήσει έρευνα ή όχι. Αυτό ζητήθηκε. Ε, από την κοινωνία των πολιτών και νομίζω ότι σε αυτόν τον κανονισμό μπορούμε να το λάβουμε περισσότερο υπόψη μας. Γι' αυτό λοιπόν σας επαναλαμβάνω θα εξετάσουμε το θέμα περισσότερο και θα καταθέσουμε βέβαια τις τροπολογίες μας. Σας ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να σας ενημερώσω ότι το σχέδιο της ε, έκθεσης ε, θα εξεταστεί στην επόμενη ε, τακτική μας συνάντηση που είναι το Μάρτιο. Πάμε τώρα στα θέματα 16 και 17. Θα τα εξετάσουμε από κοινού το 16 και το 17. Και τα δύο θέματα αφορούν στην ε, συμφωνία που προβλέπει η σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Κεντρικής Αμερικής ε, αφετέρου. Ο κύριος Παύλος Σάλμπα είναι ο εισηγητής. Θα εξετάσουμε τον εμπορικό πυλώνα αυτής της ε, συμφωνίας Και επίση ε, θα εξετάσουμε και τρίτρα ασφαλεία για την ίδια συμφωνία και για το δεύτερο εισηγητή έχουμε τον κύριο Γιώργν Λάιχτφριντ. Η εμπορική συμφωνία με την ε, Κεντρική Αμερική ε, δεν είναι τόσο επίμαχη όσο αυτή που συζητήσαμε χτες για την Κολομβία και το Περού. Και η ρήτρα ασφαλείας, όσον αφορά τη ρήτρα ασφαλείας, αυτή που ισχύει για την Κολομβία και το Περού ισχύει και εδώ για αυτή την περίπτωση, την Κεντρική Αμερική. Όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε υπάρχει διαφωνία ως προς τη διαδικασία για την ε, συμφωνία. Πρόκειται για τη Συμφωνία ε, Ελεύθερων Εμπορικών Αντολιγών που εντάσσεται στις γενικότερες συμφωνίες με την Κεντρική Αμερική ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ε, θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε με αυτή την ε, συμφωνία εμπορικών ανταλλαγών. Γιατί όπως σας είπα αφορά τη γενικότερη συμφωνία με την Κεντρική Αμερική. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους εισηγητές Ξεκινάω με τον κύριο Παύλο Σάλβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για μια τεράστια σημασία συμφωνία τόσο στο εμπορικό σκέλος όσο και στο πολιτικό και για τις δύο περιοχές. Είναι η πρώτη ε, συμφωνία ε, με περιφέρεια που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα στείλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ γρήγορα την, ε, το τελικό σχήμα και θα ήθελα να ήξερα κατά πόσο θα εφαρμοστεί το άρθρο 51 ή όχι. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τον ε, Πρόεδρο για τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί πιστεύω ότι νομικά έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά και όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, τον ευχαριστώ. Και στο κάτω-κάτω δεν θα είναι επειδή δεν έχουμε αρκετά πολιτικά επιχειρήματα. Πάντω υπάρχει μεγάλο εμπορικό δυναμικό στη συμφωνία αυτή και για τις δύο περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τώρα το 33% από το 2006 μέχρι το 2010 αύξηση των εισαγωγών. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εμπορικές συναλλαγές της τάξης του 32% δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατασκευαστικά προϊόντα τα εξάγει στη Λατινική Αμερική. Ελπίζουμε η συμφωνία αυτή, άπαξ και αρχίσει να ισχύει, θα διαφοροποιήσει κάπως τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και των δύο περιοχών. Για την Ευρώπη αυτό σημαίνει μεγάλη ευκαιρία για τις υπηρεσίες μας θα αναπτυχθεί πολύ στη Λατινική Αμερική και θα βοηθήσει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Είναι μια τεράστια ευκαιρία που μας δίνεται για επενδύσεις σε τομείς ε, με μεγάλο δυναμικό όπως είναι ο τουρισμός. Χρειάζεται φυσικά ποιότητα, ε, σωστές ε, εμπορικές τεχνικές και προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπογραμμίζουμε εδώ επίσης και ότι όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτή για τη Λατινική Αμερική στον τομέα των ονόσιμων πηγών ενέργειας, στον τομέα των υποδομών. Ξέρουμε τι γίνεται στη διόρυγα του Παναμά και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ε, πετύχουμε και να επικυρώσουμε τη συμφωνία αυτή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρόεδρο, όπως ε, γνωρίζετε, είμαι και εισηγητής για την ρήτρα διασφάλισης. Εδώ θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ρήτρα διασφάλισης η οποία να είναι αποτελεσματική και να είναι και μια ρήτρα η οποία να τίθεται εύκολα σε εφαρμογή. Ακριβώς γι' αυτό θα ακούσουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί όλος ιδιαιτέρως με το θέμα της μπανάνας. Θέλω όμω να εκφράσω και την ανησυχία μου κάπω για την επικύρωση από πλευρά των χωρών τη Κεντρική Αμερική. Ξέρετε ότι άπαξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επικυρώσει τη συμφωνία αυτή, θα αρχίσει να ισχύει εφόσον όλε οι χώρε τη Κεντρική Αμερική θα την έχουν ε, υπογράψει. Αλλά αν υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ε, από την πρώτη υπογραφή μέχρι τις επόμενες, καταλαβαίνετε ότι η πρώτη χώρα θα έχει ένα μεγάλο πλονέκτημα, γιατί το σύστημα ποσοστώσεων θα αρχίσει να λειτουργεί, οπότε οι χώρες Κεντρικής Αμερικής οι οποίες θα προστίθενται, θα έχουν λιγότερες δυνατότητες εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη επικύρωση θα υπάρχει δασμολογικό πλεονέκτημα που μπορεί να οδηγήσει με τη σειρά του σε κάποια στρέβλωση στο εμπόριο. Γι' αυτό και ενθαρρύνω τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών και το λέω μέσω των πρέσβεών τους, να φροντίσουν η επικύρωση από αυτούς να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα και ή δυνατόν ταυτόχρονα. Θέλω επίση να υπογραμμίσω ότι αυτή τη βδομάδα είχαμε μια συνάντηση με όλους τους πρέσβεις ε, της Κεντρικής Αμερικής με τους οποίους ανταλλάξαμε απόψεις για τα θέματα αυτά. Τον ε, Μάρτιο θα οργανώσουμε εδώ η Επιτροπή μας μία κρόαση κατά τη διάρκεια της οποίας θα ακούσουμε τους κύριους φορείς της οικονομίας της Κεντρικής Αμερικής, επιχειρηματίες, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κλπ. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας προκειμένου ό,τι θέλετε ε, να σας απαντήσω. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη συμφωνία αυτή λοιπόν όντω θα υπάρξει ακρόαση η οποία προβλέπεται για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, τη ΣΥΝΤΑ δηλαδή, μέσα στο Μάρτιο. Ωραία, περνάμε στην ρήτρα διασφάλισης. Η συγητής είναι ο κύριος Λίχφριτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αρκετά εύκολο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αν ε, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν παρεμφερεί προβλήματα, δεν ξέρω, οι συνάδελφοι που με το Περού και την Κολομβία μπορούν ίσως να μας ε, βοηθήσουν. Προσπαθούμε τέλος πάντων και σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όπως και στην περίπτωση της ρήτρα ε, σε σχέση με το Περού και την Κολομβία, έτσι και εδώ τίθενται κάποια συναφή ζητήματα. Και μπορούμε να αναρωτηθούμε για τα εξής. Η βιομηχανία λέμε ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει καλύτερα σε εξελίξεις που ενδεχομένως θα την πλήξουν και γι' αυτό το λόγο Κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια ρήτρα διασφάλισης ε, μοιάζει, όπως είπε και ο κύριος Μίλλερ, ο εκπρόσωπος της με μια ζώνη ασφαλείας. Ε, ε, η ζώνη ασφαλείας φυσικά, καταλαβαίνετε, δεν πουλώνει τα τραύματα, οπότε πρέπει να προσέξουμε και να έχουμε όλα τα πετούμενα μέσα στη διάθεσή μας. Όχι μόνο αυτό όμως, ενδεχομένως να χρειαστεί και κάτι άλλο. Ίσως να μην χρειάζεται η βιομηχανία να καλέσει ε, σε δράση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω οι κοινωνικοί εταίροι θα έπρεπε να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο και από τις δύο πλευρές της βιομηχανίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα και ενδεχομένω αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δυστυχώς θα πρέπει να συμφωνήσω και με τον κύριο ε, Στέρντι δηλαδή είπε ότι ίσως χρειαζόμαστε ένα τρόπο να βοηθήσουμε όσους έχουν προβλήματα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανάπτυξη. Εγώ θα ήθελα λοιπόν από αυτού να ρωτήσω το εξής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτή τη ρήτρα ε, θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να ενισχύσουμε παραγωγούς ε, που παράγουν ε, προϊόντα βιολογικής ε, καλλιέργειας ή δίκαιου εμπορίου, κυρίως στον τομέα της μπανάνας. Γνωρίζουμε ότι το fair trade, το θεμητό εμπόριο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στον τομέα της ε, μπανάνας, ε, ούτε και η βιολογική καλλιέργεια είναι τόσο συχνή στην παραγωγή μπανάνας ε, όσο θα έπρεπε να είναι, εν πάση περίπτωση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το εξής. Δεν... Είμαι εισηγητή και επίση κοιόδη εισηγητή για τη συνολικότερη συμφωνία. Οπότε βοήθησε λίγο τον κύριο Σάλβα για αυτό το θέμα. Α προσθέσω και το εξή. Είναι προφανέ ότι για μια ρήτρα διασφάλιση το κοινωνικό θεματολογία, οι κοινωνικοί στόχοι δεν έχουν ε, μια α το πω κατοχυρωμένη θέση. Τέλο πάντων, αληθεύει αυτό, είτε συμφωνώ εγώ είτε όχι. θα πρέπει να ασχοληθούμε όχι μόνο με τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, με στόχο όχι μόνο να βοηθήσουμε τον πληθυσμό στην Κεντρική Αμερική, αλλά για να αυτό βοηθηθούμε, διότι υποφελούμαστε κι εμεί από την ανάπτυξη ε, από μια πιο ευημερούσα και ασφαλέστερη οικονομία στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, διότι ενδέχεται να αυξηθούν οι εξαγωγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, άρα θα είναι αμοιβαία υποφελέ τελικά το νέο σύστημα. είδου αυτά ήθελα χονδρικά να σας εκθέσω σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, με μεγάλη χαρά θα επεξεργαστώ οποιασδήποτε προτάσεις θέλετε να υποβάλλετε. Ε, κοίταξα τις τροπολογίες ε, της Επιτροπής Γεωργίας Εντάχη, χτες δηλαδή, και θα έλεγα ότι είναι εύστοχες ε, ως επιτοπλίστων οι τροπολογίες. Για το θέμα της μπανάνας δεν νομίζω να μου δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα οι τροπολογίες. Σας ευχαριστώ για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Αν έχετε προτάσεις, συστάσεις, οτιδήποτε, θα είμαι στη διάθεσή σας, θα σας βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λάιχτφριντ. Όπως είπε ο Γκαμπρίλ Μάτο προηγουμένως, σχετικά με τον κανονισμό περί ρητρών διασφάλισης ε, για την Κολομβία και το Περού. Τα ίδια λοιπόν περίπου ισχύουν και με αυτή τη συμφωνία. Μήπως θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ή... ή να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά που είπατε προηγουμένως ισχύουν και για αυτή τη συμφωνία. Όχι, όντως ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Μόνο ευχαριστώ πολύ, τίποτα άλλο. Ωραία, ευχαριστούμε κι εμείς. Οπότε τώρα συζήτηση. Θέλει κανείς το λόγο, η Σκιώδης, δεν σου λέω εδώ. Α, όχι, ο κύριος ε, Σολτς είναι εδώ. Η πράσινη μετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον, στους συζητητές για τη δουλειά που έχουν κάνει. Όντω αυτό είναι το μαγικό με τι διαπραγματεύσει. ότι τελικά αντιστρέφονται οι καταστάσει πλήρω μερικέ φορέ στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Όλοι οι υπουργοί τη Κεντρική Αμερική είχαν κλείσει την πόρτα πίσω του, μετά από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέλει να επιβάλλει γαλακτοκομικές ποσοστώσεις και μια εβδομάδα μετά άλλαξαν, δεν ξέρω, κάποιος ίσως μας πει κάποια μέρα τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε σε αυτή τη συμφωνία. Έχω να σχολιάσω λίγο κάποια σημεία που για μένα έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα των υπέρ και των ε, κατά, αλλά και με την περιφερειακή ολοκλήρωση. Ο συνάδελφος πριν είπε κάτι πολύ σημαντικό για αυτό το τελευταίο. Όντως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εφόσον οι ποσοστώσεις δεν κατανέμονται συλλογικά, όταν δηλαδή έχουν επικυρώσει όλες οι χώρες, γιατί τότε αμφισβητείται μία περιφερειακή μονάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι απόλυτη για το ότι οι ποσοστώσεις θα κατανεμηθούν δίκαια με τον ίδιο τρόπο μεταξύ όλων των χωρών που θα έχουν επικυρώσει τη συμφωνία. Το δεύτερο που έχω να σχολιάσω είναι το εξή. Ποιο θα υποφεληθεί από τη συμφωνία αυτή τελικά και ποιοι είναι οι τομεί εκείνοι οι οποίοι πλήττονται περισσότερο. Α δούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τον δημοσιονομικό τομέα. Αυτά που έλεγε η μελέτη αξιολόγησης είναι ότι οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής χάνουν περίπου πλήρως τον έλεγχο του κλάδου των, τραπεζικών, των τραπεζών και, των, ε, ασφα... και Πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να περάσετε έτσι. Εγώ δεν νομίζω. Γιατί ακόμα και αν βάλουμε στην πάντα τον Παναμά που ξέρουμε ότι είναι δημοσιονομικός παράδεισος. Το ίδιο ισχύει και για διάφορους μηχανισμούς οι οποίοι τίθεται υπό αμφισβήτηση. Δεν είναι σημαντικό για την Κεντρική Αμερική να κρατήσει ένα χώρο ε, δημόσιας πολιτικής, είτε πρόκειται για την πολιτική της στήριξη των νέων επιχειρήσεων, είτε για κάτι άλλο. Και όμως χάνουν όλο και περισσότερο περιθώριο οι χώρες αυτές προκειμένου να φτιάξουν τα πράγματα όπως θέλουν για την ανάπτυξή τους και ε, κερδίζουν οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Για τους πράσινους λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση αλλά επιμονή μου βάσεως να συζητάμε και να βλέπουμε το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει σε αυτές τις ε, ε, συμφωνίες. Εμένα δεν με ικανοποιεί το να μου πείτε «Α, θα προβλέψουμε αντισταθμίσματα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς». Έχουμε το Ταμείο για τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση. Το ότι όμως βάζουμε δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτούμε τους αγρότες μας οι οποίοι θα εξαφανιστούν, για μένα δεν είναι ένας έξυπνος τρόπος να αντιμετωπίζουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και συμφωνώ με τις ε, παρατηρήσεις του προελίσαντος ε, όσον αφορά γενικά αυτόν τον κανονισμό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο εισηγητές για το γεγονός ότι όρισαν την κατάσταση και επίσης ε, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και για το γεγονός ε, ότι έλαβαν υπόψη τους ε, τις γεωργικές εξελίξεις. Θα ήθελα λοιπόν να φέρω δύο πράγματα. Στη συζήτηση που ανέφερε ο κύριος Άλμπα, τη συζήτηση την οποία είχαμε με τους πρέσβεις, Εκεί αναφερθήκαμε στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν επενδύσεις. Επενδύσεις ε, στις χώρες αυτές ε, εφόσον αυτές επιθυμούν ε, την οικονομική τους ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτό αφορά και τα κεφάλαια της συμφωνίας ε, που έχουν σχέση με τα χρηματοοικονομικά. Όμως αυτά ε, κατά κάποιον τρόπο υπολείπονται κυρίως διότι οι διεθνείς ε, τράπεζες εξακολουθούν να κατησχύουν στον οικονομικό τομέα ε, της Κεντρικής ε, Αμερικής. Υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη χρηματοπιστωτική δομή. Είναι οι τράπεζες εκείνες ε, οι οποίες και λόγω της κρίσης στην Ευρώπη υπερισχύουν όπως σας είπα και γι' αυτό αντιρωτάται κανείς κατά πόσον πράγματι ε, υπάρχει επιθυμία για ε, περιφερειακή ανεξαρτησία. Αυτή, αυτό ισχύει αν θέλετε στο Ελσαλβαντόρ, στις ε, Ονδούρες, στη Νικαράγουα. Είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ε, κυρίως όσον αφορά ε, στα εργατικά δικαιώματα, στην ε, εξέλιξη των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας, έτσι ώστε να προκύψει οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό το προσμένουν σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε. Το δεύτερο που πολύ σωστά ετέθη είναι ποιος θα ωφεληθεί από τη συμφωνία. Και νομίζω ότι στην ακρόαση που θα ακολουθήσει θα πρέπει να διερωτηθούμε, να δούμε λιγάκι ε, πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις ε, διατάξεις ε, της συμφωνίας. Και εδώ επανέρχομαι στην χθεσινή ακρόαση. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις δύο όχτες του Ατλαντικού και στην Ευρώπη και στην Αμερική θέλουμε να βοηθήσουμε ε, βεβαίως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κεντρική Αμερική. Αυτά είχα καταρχήν να σας πω και νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι η εργασία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία. Πρόεδρος, Ας ακούσουμε τώρα την ε, Κομισιόν ε, σχετικά με την εμπορική συμφωνία ο κύριος Ματίας Γιώργενσεν και για την ρήτρα ασφαλείας ο κύριος Φεντρίχ Μισελ. Ο κύριος Γιώργενσεν παρακαλώ ξεκινάει. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ε, ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Κάποια σύντομα σχόλια έχω μόνο και θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τι παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής σας. Πρώτον, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τη συμφωνία αυτή και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα περατώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες ούτω ώστε η θέση σε ισχύ να λάβει χώρα το ταχύτερο δυνατόν. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία θα έχει θετικό αντίκτυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υψηλής ποιότητας εξάλλου και μας προσφέρει πρόσβαση σε αγορέ που μα ενδιαφέρουν. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία είναι εξίσου υποφελής και για την Κεντρική Αμερική, διότι χάρη σε αυτή οι χώρες ε, της Κεντρικής Αμερικής θα έχουν τη δυνατότητα να ε, αποκτήσουν επιπρόσθετες εξαγωγικές δυνατότητες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να τονώσουν την ανάπτυξή τους, θα μπορέσουν να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους και τις εξαγωγές τους προς την Ένωση. Το τρίτο και επίσης βασικό είναι το εξής. Η συμφωνία αυτή ευθυγραμμίζεται κατά τη γνώμη μας, σε μεγάλο βαθμό με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει εν γένεια η Ένωση για την Κεντρική Αμερική. Περιφερειακή δηλαδή ολοκλήρωση και εξάλληψη της φτώχειας. Είναι μια συμφωνία από περιφέρεια σε περιφέρεια, από περιοχή σε περιοχή, region to region ε, και αποσκοπούμε, όπως είπαμε, στην περιφερειακή ανάπτυξη τη Κεντρική Αμερική από τι αρχέ δεκαετία του 80 και τη στήριξη τη ειρηνευτική διαδικασία ε, επί τόπου. Έχουμε στενή σχέση με αυτέ τι χώρε. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντική συμβολή σε αυτό. Να σα ε, παρουσιάσουμε την κατάσταση. Πού έχουμε φτάσει στη διαδικασία. Έχουμε καταθέσει πρόταση ε, προ υπογραφή από το Συμβούλιο τη Συμφωνία τον Οκτώβρη. Βαίνουν εσύ οι εργασίε του Συμβουλίου και μάθαμε ότι αναμένεται στο Συμβούλιο η απόφαση για την υπογραφή να έχει ληφθεί κατά το μήνα Μάιο και στη συνέχεια θα προβούν στην ε, υπογραφή με τους εταίρους της Κεντρικής Αμερικής ε, ε, το ταχύτερο δυνατόν, ευελπιστούμε μέσα στον Ιούνιο κατά τα μέσα Ιουνίου. Στη συνέχεια το Συμβούλιο θα διαβιβάσει την επίσημη συμφωνία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σύμφωνη γνώμη. Μετά την υπογραφή λοιπόν θα λάβει επίσημα το σχέδιο συμφωνίας, μάλλον τη συμφωνία, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ καλό που ήδη αρχίσατε να την επεξεργάζεστε. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω κάποια επιμέρους ζητήματα. Πόσο στόσεις. Ε, το θέμα δηλαδή αν ε, είναι ισότιμη η κατανομή των ποσοστώσεων σε όλες τις χώρες ε, της Κεντρικής Αμερικής. Εμείς συμφωνήσαμε για περιφερειακές ποσοστώσεις στην Κεντρική Αμερική και τους αφήσαμε τη δυνατότητα εκείνοι να αποφασίσουν την κατανομή για τη ζάχαρη, για το ρύζι σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Εκείνες θα αποφασίσουν και κατά τη γνώμη μας ε, αυτό θα τονώσει, θα ενισχύσει την περιφερειακή ολοκλήρωση που επιθυμούμε. Έχουμε επίσης ένα αρκετά πλούσιο κεφάλαιο για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στη συμφωνία. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες από αυτού, αλλά όπως γνωρίζετε, το ίδιο συνέβη και σε περίπτωση σε, ως προς άλλες συμφωνίες. Δηλαδή, οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν δεσμεύσει για όλα τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφεντέρου χώρες της Κεντρικής Αμερικής, ως προς την ε, υλοποίηση και την ουσιαστική τήρηση ε, των ε, βασικών εργασιακών δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνται στις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, επίσης ε, προβλέπεται μηχανισμός ε, διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών και ένας ειδικό μηχανισμός επίλυσης των διαφορών ή εξέτασης αμφιλεγόμενων ζητημάτων για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Σφαιρικά κρίνουμε ότι είναι ικανοποιητική η συμφωνία και ελπίζουμε να τύχει ευρύτατη υποστήριξη στο Κοινοβούλιο, διότι θεωρούμε ότι Μέσω αυτή τη συμφωνίας θα περάσουμε ένα σημαντικότατο μήνυμα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη που προσφέρουμε στην Κεντρική Αμερική, διότι ας ε, συνυπολογίσουμε ότι βιώνουν μια σχετικά δύσκολη περίοδο και το χρειάζονται. Θέλουν να δουν ότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστική και η ταχύτητα θέση σε ισχύ είναι και το ιδανικότερο μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε. Πρόεδρος, Έχουμε και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου για την ε, λήψη απόφαση για αυτή τη συμφωνία. Φυσικά δεν μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία πρωτού επιληφθεί επίσημα το Κοινοβούλιο του ζητήματος με την υποβολή της ε, υπογεγραμμένης συμφωνίας ε, σχετικά ε, με τον μηχανισμό διασφάλισης. Ποιος θα μιλήσει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το θέμα αυτό είναι το κατά πόσο θα χρησιμοποιήσουμε για τα βιολογικά προϊόντα τη ρήτρα αυτή διασφάλισης. Πρόκειται για κάτι ουδέτερο. Το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρξει μεγάλη αύξηση ή όχι και τι μέσα, δηλαδή, και τι μέσα θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την περίπτωση. Τώρα για, την, για το μηχανισμό σταθεροποίησης για την μπανάνα δεν πρέπει να μιλάμε για ποσοστώσεις εδώ μιλάμε για όγκους ενεργοποίησης και όχι για ποσοστώσεις, γιατί οι ποσοστώσεις καταργήθηκαν ως υποχρέωση από πλευράς του ΠΟΕ και χρησιμοποιούμε ένα δεσμολογικό σύστημα μόνο για την μπανάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άλλες παρατηρήσεις, εισηγητές μήπως, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, το πρώτο που έχω να πω στους εισηγητές, ιδιαίτερα στο Γιάνν είναι ότι η συμφωνία αυτή όντως πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή ολοκλήρωση στην Κεντρική Αμερική. Ελπίζουμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαρίστως να συζητήσω μαζί σας για το θέμα της κατανομής των ποσοστώσεων και πολύ χαίρομαι που ακούω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα. Άρα θα το συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση. Για το οικονομικό σύστημα τώρα, το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα είναι βέβαια πιο ανταγωνιστικό από εκείνο της Κεντρικής Αμερικής. Άρα λοιπόν ε, προβλέπεται ε, μεγαλύτερη παρουσία των δικών μας τραπεζών στην Κεντρική Αμερική. Δεν, μπορούμε, δεν θέλουμε να την αποφύγουμε την παρουσία αυτή, αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι η παρουσία μας εκεί να οδηγήσει σε ένα οικονομικό σύστημα πιο ανταγωνιστικό και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες οι κεντροαμερικανικές επιχειρήσεις μέσω περισσότερου ρευστού για να δράσουν. Αυτή, αυτός πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου ο στόχος μας. Τώρα ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Είμαι πεπισμένο όπως και η Επιτροπή, ότι με τη συμφωνία αυτή κερδίζει και η Κεντρική Αμερική και η Ευρώπη. Αυτό φαίνεται και από τη μελέτη του London School of Economics που προβλέπεται αργότερα σήμερα. Ε, θα μπορέσουμε να δούμε έτσι τα πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ για τον κανονισμό ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι ε, μας έδωσε τροφή για σκέψη, κυρίως ε, όσον αφορά ε, στα βιολογικά προϊόντα και το θεμητό εμπόριο. Θα χρησιμοποιήσω το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας για να δω λιγάκι αν μπορώ να αλλάξω το πνεύμα που χαρακτηρίζει αυτή την ρήτρα. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε την ε, απόφαση του ε, Συμβουλίου. Τώρα, ε, Φτάσαμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ να προετοιμάσετε τις κάρτες σας και τον κατάλογο ψηφοφορίας.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 Λοιπόν, ε, δεν θα ψηφίσουμε τώρα για την έκθεση της κυρίας Μαριέλ Ντεσαρνέσε, για την έκθεσή της, εκείνη το ζήτησε εξάλλου χθες. Θα περάσουμε λοιπόν ε, απευθείας στην έκθεση του κυρίου Φιέλνερ για το GSP, το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων. Θέλει ο εισηγητής το λόγο, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομο, ε, Πρόεδρε. Δράτω με τι ευκαιρίε για να ευχαριστήσω όλου όσου ενεπλάκησαν ε, στην εκπόνηση τη πρόταση. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Πάρα πολλέ τεχνικέ τροπολογίε μα απασχόλησαν και θα ήθελα τουλάχιστον να, να ευχαριστήσω την ε, Ελένα από την Γραμματεία γιατί με υποστήριξε με εκπληκτικό τρόπο και δεν ήταν και η μόνη. Πριν αρχίσουμε λοιπόν ευχαριστώ προς όλους. Πρόεδρος για να έχουμε σαφή ε, εικόνα της πολυπλοκότητας. Έχουμε 24 ε, τροπολογίες από τον εισηγητή, 182 από τα μέλη της Επιτροπής, 20 από την Επιτροπή Ανάπτυξης και διάφορες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που ελπίζω να διευκολύνουν τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ευχαριστούμε και εμείς τον εισηγητή. Εργαστήκατε με εξαιρετικό τρόπο και σας ευχαριστούμε που συνεργαστήκατε με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, κυρίως με τους σκιώδεις εισηγητές. Κατόπιν τούτου, ας προχωρήσουμε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε ομού. Block vote όπως βλέπετε. Υπαριθμών 1. Υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της Επιτροπής Ανάπτυξη. Υπέρ παρακαλώ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. 46, 47, 48 και 59 το πρώτο τμήμα. Είναι όλες ταυτόσιμες. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογίες 51 54, 55, 56, 57 και 59 δεύτερο τμήμα. Ταυτόσιμες επίσης. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε πάλι για τις τροπολογίες 51 και ακόλουθες μέχρι την 59 δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ. Άρχεται. Πέραση ψηφοφορίας. Απερίφθησαν όντως. 52 και εφεξής είναι ταυτόσιμες, υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές απορρίπτονται επίσης. Τροπολογία 61. Συζητά, συγγνώμη, ο Πρόεδρος διορθώνει. Οι 60 και 5 ταυτόσημες ψηφίζουμε, υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτονται. Αυτή τη φορά θα το πω σωστά. Η 61 υπέρ. Κάτα. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. 66 πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 68, η 70 και όλες μέχρι το 73. Όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος. Μέχρι την 73. Τρεις τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 66, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα θα περάσουμε στις 80 και 84. Είναι ταυτόσιμες και πάλι. Υπέρ παρακαλώ. Μάριο Δεβίδο, δεν ναι, υπερψηφίζει τη δική σου την τροπολογία. Τι γίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 τώρα. Υπέρ. Κατά απορχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φτάνουμε στη συμβιβαστική υπαριθμών 2 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 92 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση, ευχαρίστως. 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Μα τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική μου κάρτα, λέει ο πρόεδρος. Δεν δουλεύει πια. Εγώ υπέρ θα ψηφίσω, προφανώς. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Δεν δουλεύει. Δουλεύει. Για την 92 ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. 93 υπέρ. Η ε, ισοψηφία ήταν 15 προς 15 ήταν η ψήφη. Με τη δική μου την ψήφο. διάφορα σχόλια εκτό μικροφώνου από τα μέλη τη Επιτροπή, Απαντάει ο πρόεδρο ότι δεν έχει γίνει καμία καταγγελία επί τη διαδικασία. και εγώ λυπάμαι, αλλά περίφθη. Τι να κάνω. 93 υπέρ. Κάτα. Αποχέ, απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κάτα. απόχέ. απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 94. 94. Α, και την 7. Μαζί θα τις ψηφίσουμε, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 τώρα υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Και η 9. Ομού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 είναι και πάλι από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102. Υπάρχει μία πρόταση για προφορική τροπολογία. Ενστάσεις υπάρχουν, μπορούμε να συμπεριλάβουμε την προφορική. Δεν βλέπω να προτάσει κάποιος ενστασή. Πολύ ωραία. Ε, αναφέρεται στον κατάλογο ψηφοφορία η προφορική τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε με αυτήν υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία μου, υπαριθμό 2, μπλοκ vote 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η 107 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίθηκε. 4 από την ΤΕΒΕ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 117 υπέρ κατά απόχες Απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 120 και 21 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Επαλήφευση για τις 120 και 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, πέρας. Όντως, όντως απεριφθεί. 122, 123 και 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 22, 23, 24, παρακαλώ. Πέρας. Όντως απερίφθησα. 15. Υπέρα. Κάτα. Άποχες. Παλήθευση. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται όντως. Η 125 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 127 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 130. Όχι, 29 διορθώνει ο πρόεδρος. 129 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 11 τώρα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 134 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβιβαστική αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 τώρα. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Παρακαλώ. Μπορείτε να ελέγξετε τι έγινε παρακαλώ με την τροπολογία 136. Μου λένε ότι καταπίπτει εξαιτία τη συμβαστική τροπολογία. Μπορούμε να το ελέγξουμε. Κύριε Φιέλμα, τι έχετε να πείτε για την 136. Καταπίπτει, όχι. Νομίζω ότι αν καταλαβαίνω έχουν αποσυρθεί άλλες. Αλλά εγώ έχω μια σολομόντια λύση. Να την ψηφίσουμε και μετά να ελέγξουμε τεχνικά αν ε, στέκει όχι. Έτσι, just in case, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, για να μην ξαναβρεθούμε και ξαναψηφίζουμε κτλ. Ωραία, ας ψηφίσουμε τότε για την 136. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. 160. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε πράγματι. Τροπολογία 18 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, α, καταπίπτει, δεν ψηφίζουμε. 23 τότε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει και για την 183 ε, που ψηφίσαμε μαζί ουσιαστικά γιατί είναι ταυτόσιμες. Αλλά και 6, 7, 8, 9 και 190. 185 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και έτσι προχωράμε και φτάνουμε σε ψηφοφορία των τροπολογιών 193, 94, 95, 96, 98 και 199 επειδή είναι ταυτόσιμες μεταξύ τους. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 201 και 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 33 λένε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. επτά τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και έτσι φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Επί της πρότασης της Επιτροπής, έτσι όπως τροποποιήθηκε αυτή, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίες. Το αποτέλεσμα είναι 22 υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές. Ε, ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 6 κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω όμως να ζητήσω από την Επιτροπή μας δύο πράγματα. Ή και τον Πρόεδρο ίσως, δεν ξέρω ποιον πρέπει να ρωτήσω. Όταν ξεκινήσουν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο για να πετύχουμε κάποια συμφωνία, πότε θα είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι σύντομα. Και θέλω επίσης να ξέρω για την επόμενη Ολομέλεια τι προβλέπετε. Πρόεδρος, έχουμε κάτι που πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα, να δούμε κατά πόσο θα προχωρήσουμε μέσω σε πρώτη ανάγνωση, σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης ή όχι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για πακέτο, δηλαδή ότι ξεκινούμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά πάμε στην επόμενη δυνατόν ολομέλεια. Ωραία, έτσι διευκρινίζεται η πρόταση. Ποιος είναι υπέρ, λοιπόν, αυτή της διαδικασίας ακριβώς. Να αρχίσουμε αμέσως τι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, δηλαδή, χωρίς βέβαια να προκαταλαμβάνονται οι ψηφοφορίε που θα γίνουν και το αποτέλεσμα δηλαδή των ψηφοφοριών που θα γίνουν στην Ολομέλεια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι διαπραγματεύσεις η διαπραγματευτική ομάδα ο ο πρόεδρος, όπως πάντα, ο Κρίστοφερ Χέλνερ που είναι εισηγητής βέβαια, e ε, η σκιώδης Δέβιτ Μάρνες, Δίν, λοιπόν ο Μαρινάλντι, Άλβερ, Λομπερστέρντι, το ECR, ε, Αντιρρήσεις. Είναι έτσι κι αλλιώς η συνήθιση διαδικασία. Καλώς θα έρθω σε επαφή μαζί σας για να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Περνάμε τώρα στο σημείο 20. Έχουμε και εδώ να ψηφίσουμε. Πρόκειται για σύμφωνη γνώμη εδώ. Όσον αφορά το τροπμένο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της Διεθνούς Ομάδας Μελετών για το Ελαστικό. Είμαι εισηγητής και λέω να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Αυτό προτείνω. Ψηφίζουμε όμως. Ε, μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά, έτσι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Έτσι φτάσαμε στη λήξη της ψηφοφορίας. Και πάμε λίγο πίσω. Πάμε στο σημείο 14. Άκτα. Αρχίσαμε χτες την ε, σχετική συζήτηση, αλλά ακούσαμε μόνο τον Επίτροπο Γι' αυτό και αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουμε σήμερα με τη συζήτηση. Λοιπόν, ποιο έχει στήσει το λόγο. Ε, όντως, ο κύριο Κάρδιτ είναι από χτες, μας έχει μείνει για τη συμφωνία αυτή. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ χτες και να ακούσω αυτά που είπε ο Επίτροπος. Αν θέλετε να μιλήσετε κι εσείς για τα υπέρ και τα κατά, έχω ολόκληρο κατάλογο, έτσι, οπότε σας βάζω και εσάς τον κατάλογο. Είναι διαδικαστικό αυτό που θέλετε να πείτε. Αν ήταν διαδικαστικό, γι' αυτό σας έδωσα το λόγο. Αλλιώς έχω ήδη κατάλογο εδώ. Δεν είχα την ευκαιρία να γραφτώ, πρόεδρε. Εντάξει, Φυσικά, όσο πιο γρήγορα πάρω το λόγο, τόσο το καλύτερο για να μπορέσω να πω και εγώ αυτά που θέλω να πω. Λοιπόν, έχω εδώ τον χθεσινό κατάλογο, όπως σας είπα. Και πρώτος από όλους είναι ο συγκητής μας, ο κύριος Ντέβιτ Μάρτιν. Έχεις το λόγο, Ντέβιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, Επίτροπο που ξανάρθε. Τον βλέπω εδώ. Ωραία. Όπως είπε λοιπόν χτες ο Επίτροπος, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίμαχο και μέσα στο Κοινοβούλιο και σε σχέση με τις εργασίες του Κοινοβουλίου μας εδώ. Πριν από δύο μέρες με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών δεχτήκαμε ε, αναφορά με 2,5 εκατομμύρια υπογραφές, πράγμα το οποίο δείχνει το εύρος του ενδιαφέροντος. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες φαντάζομαι ότι θα έρθω σε επαφή και μόνο γίνεται περισσότερο εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να κατανοήσω τις ανησυχίες τους και για να συμμεριστώ μαζί σας τις ανησυχίες τους αυτές. Θα αρχίσω λοιπόν με το θέμα με το οποίο ξεκίνησε και χτες ο Επίτροπος, το θέμα της διαφάνειας. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν εμπιστετεύεται ο κόσμος στην άκτα είναι εξαιτία του τρόπου με τον οποίο έγινε διαπραγμάτευση. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εκείνων που διαπραγματεύονται και εμείς ως Επιτροπή Εμπορίου καταλαβαίνουμε ότι η ισορροπία να είναι δηλαδή ελαστική η κατάσταση αλλά συγχρόνως ε, να υπάρχει διαφάνεια, να στο ότι έπρεπε να γίνει και κλεισμένον των θυρών. Αλλά τελικά το απόρριτο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση για μας δεν ε, είναι κάτι που θέλαμε. Είχαμε ψηφίσματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκφράσαμε τις ανησυχίες μας, ε, υιοθετήσαμε και κείμενα με τα οποία ζητούσαμε μεγαλύτερη διαφάνεια, να είμαστε πιο ανοιχτοί όσον αφορά τις διαπραγματεύσει ε, για το ΑΚΤΑ. Πρέπει επίσης να πω ότι πολύ συχνά Ακούγαμε ότι η κοινωνία των πολιτών δεν είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή μαζί μας, για παράδειγμα. Υπάρχουν δηλαδή απόλυτα θεμητές ανησυχίες για τον τρόπο που έγινε η διαπραγμάτευση για το ΑΚΤΑ. Όμως ό,τι έγινε, έγινε. Και το κοινοβούλιο μας καλείται να αποφανθεί βάσει του κειμένου που έχει στη διάθεσή του. Επιτρέψτε μου όμως να μπει στα πρακτικά αυτό ότι ε, πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή ε, ε, πνευματική ιδιοκτησία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ξέρουμε ότι πρόκειται στο κάτω-κάτω για την πρώτη ύλη για την επιτυχία της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αλλιώς στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια σκηνή. Και δεν πρόκειται μόνο για τα οικονομικά συμφέροντά μας τώρα υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να αποβούν ε, επικίνδυνα αν δεν προστατεύσουμε ας πούμε τα φάρμακα ή ακόμη και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Όπως και να έχει πάντως το πράγμα. Δεν λέω ότι επίτηδε προσπαθεί άκτα να το κάνει αυτό, αλλά κατά λάθο μα το κάνει. Γιατί ξέρετε, εμεί λέμε ότι ο διάβολο βρίσκεται στι λεπτομέρειε. Και η ανησυχία μου είναι ακριβώ αυτή, ότι δεν έχουμε εδώ λεπτομέρειε. Βλέπουμε το κείμενο, αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από τι γραμμέ του κειμένου. Γι' αυτό και οι ανησυχίε μου έχουν να κάνουν περισσότερο με το πώ θα ερμηνευτεί το κείμενο και πώ θα τεθεί σε εφαρμογή. Ο Επίτροπος πολύ σωστά αναφέρθηκε σε πράγματα που λείπουν εγώ. Αυτό που θέλω είναι να συζητήσω βάσει γεγονότων. Είναι σωστό να πούμε ότι δεν υπάρχει το three strikes rule στο κείμενο αυτό. Ότι δηλαδή μετά από τρεις παραβιάσεις υπάρχουν κυρώσεις είναι στο σχέδιο που διαπραγματευτήκαμε, δεν βρήκαμε αρκετά πράγματα. Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, δεν υπάρχει μνήμα στο κείμενο της άκτα όσον αφορά τα άτομα. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξέρω αν σε ένα MP3 έχει κάποιος φορτώσει κάτι νόμο ή παράνομο, ξέρετε πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά πώς θα το εντοπίσουμε. Δεν αποτελεί αυτό μέρος της διαδικασίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δεν ξέρουμε πώς οι διάφοροι φορείς του διαδικτύου θα ερμηνεύσουν αυτά που αναφέρονται στη συμφωνία. Οι φόβοι μας δεν έχουν να κάνουν με αυτό που αναφέρεται στο κείμενο για τα, τις υποχρώσεις που έχει κανείς. Ωραία, οι υποχρεώσεις που μιλάνε για τον έλεγχο κτλ. Το θέμα τι είναι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να... Ε, το ότι λέει ότι πρέπει να σταματάμε κάποιον να διαπιστωθεί ότι προσπαθεί κάτι να κατεβάσει. Πώς ερμηνεύεται αυτό τελικά. Η συμφωνία, και μας το επιθυμίζει ο Επίτροπος, έχει να κάνει για τις αντιγραφές που γίνονται για λόγους εμπορικούς. Και μπορεί να πει ότι υπάρχει και προηγούμενο που να μιλάει για την εμπορική χρήση του copyright. Όμως αν δεν είσαι εμπειρογνώμονας, αν ε, είσαι ένας αξιωματούχος, είτε ε, συνοριοφύλακας, πώς θα το καταλάβεις αυτό, πώς ορίζεται η εμπορική αυτή χρήση στην ε, Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός, χρειαζόμαστε όμως σαφήνεια για το πώς θα τεθεί σε εφαρμογή και τι σημαίνει σε εμπορική κλίμακα, πώς ερμηνεύεται αυτό. Τώρα για τα γενώσιμα φάρμακα, τα αντίγραφα. Εδώ πάλι υπάρχει διάσταση. Απ' τη μια, εντάξει, καταλαβαίνω, λέει ότι η πατέντα δεν καλύπτεται από την άκρη του Επίτροπος. Τα γεννόσιμα φάρμακα δεν καθίστανται παράνομα από τη Συμφωνία Άκτα. Ναι, αλλά και πάλι, οι σενάριοφύλακες τι θα κάνουν, πώς θα ενημερώσουν ε, την αστυνομία και πότε. Ξέρουμε από παρελθούς εμπειρία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ότι τα γενώσιμα φάρμακα κατάσχονται πολλές φορές παράνομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, έχει την υποχρέωση όταν πρόκειται για παραπημένα προϊόντα να τα κατάσχει στα σύνορα. Αλλά βλέπετε ότι εδώ ακόμα και όταν δεν πρόκειται για θέμα copyright, τα γενώσιμα κατατάσσονται συχνά με, μαζί με τα πρωτότυπα γιατί έχουν την ίδια σήμανση. Γιατί τα γιατροί, τα νοσοκομεία αναγνωρίζουν τις ουσίες τα φάρμακα αυτά. Κάποιος όμως μπορεί να νομίζει ότι πρόκειται για ε, παραποίηση φαρμάκου. Και μήπως με την ύπαρξη της άκτα τώρα κινδυνεύουν να υπάρξουν τέτοιες παρεξηγήσεις στα σύνορα και κατασχέσεις οι οποίες θέτα και σε βάρος του αναπτυσσόμενου κόσμου αλλά και των δικών μας υπηρεσιών. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα που τίθενται. Η Επίτροπος βέβαια μπορεί να μου πει μα κύριε Μάρτιν. Τώρα εδώ ε, γίνεται ανησυχίε που δεν έχουν κανένα νόημα. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ. Θέλω να είναι πιο σαφή η συμφωνία αυτή η άκτα, να γίνει, να καταστεί πιο ξεκάθαρη μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να μπορεί και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με αυτή. Σε μια συνέντευξη τύπου πριν από δύο μέρες είπα ότι ε, απατύχημα βρέθηκα να είμαι εισηγητής. Όπως ξέρουν και οι συνάδελφοι, συνήθως κάποιος επειδή ενδιαφέρεται να λαμβάνει μια έκθεση. Εδώ όμως, από την άλλη μεριά μπορεί να είμαι και ο τέλειος, όχι εξαιτία των δικών μου ε, ικανοτήτων, αλλά επειδή έρχομαι με ανοιχτό πνεύμα και δεν έχω προκαταλήψεις, δηλαδή δεν έχω αποφασίσει από πριν, δεν ξέρω από πριν ε, ποια ε, πρέπει να είναι η θέση μας. Έτσι ξεκίνησα. Ξέρω ότι η Επιτροπή θέλει να αναμειχθεί και το δικαστήριο. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποβάλει τις δικές του ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δούμε κατά πόσο η συμφωνία αυτή είναι συμβατή με τις συνθήκες και κατά πόσο είναι και συμβατή με τη Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Δεν ξέρουμε κατά πόσο το δικαστήριο θα έχει απαντήσεις, αλλά θέλω να ξέρω επίσης αν είναι συμβατή η συμφωνία αυτή με τις διεθνείς μας συμφωνίες ή με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Αν θα είναι κάτι θετικό τελικά. Το δικαστήριο Ελπίζω να μπορέσει να μου απαντήσει στις ερωτήσεις αυτής. Επίσης, όπως σας είπα και πριν, πιστεύω ότι ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή η άκτα. Γι' αυτό και έχω να προτείνω το εξή στην Επιτροπή μας. Να χρησιμοποιήσουμε το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, αλλά να μην ετοιμάσουμε τελική έκθεση, αλλά μια προσωρινή έκθεση. Μια προσωρινή βάσει της οποίας θα μας ε, γνωμοδοτήσουν οι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και θα έχουμε και τις απαντήσεις μας έτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη στην ιστοσελίδα υπάρχει ένα αλλά δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Αυτό που θέλω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, για παράδειγμα, να μας πει, όχι απλώς να μας πει, να μας διαβεβαιώσει, για το τι οδηγίες, τι αιτήσει, τι συμβουλές έχει ζητήσει, θα ζητήσει για να δούμε πώς τελικά θα τεθεί σε εφαρμογή η άκτα. Να δούμε τι κατευθυντήρες γραμμές θα δοθούν στις υπηρεσίες ε, παρόχους ε, διαδικτύου για να ξέρω τελικά ποια είναι τα δικαιώματα των μεν και ποια των δε, των χρηστών. Θέλω επίσης να ξέρω με κάθε λεπτομέρεια πώς θα τεθεί σε εφαρμογή άκτα και τις ερωτήσεις μας δεν πρέπει να τις κάνουμε μόνο στην Επιτροπή αλλά και στις χώρες μέλη. Χέλτη ειλικρινά με εξέπληξε όταν ο Βουλγαρός ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα ήταν έτοιμος να εφαρμόσει την άκτα που θα, διακρίνει, που θα κάνει διακρίση βάρος των πολιτών. Τώρα ίσως δεν κατάλαβε ότι είναι ο μόνος γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει ποινές γιατί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία και ακριβώς γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουν οι χώρες μέλη. Θα ήθελα δηλαδή και οι χώρες μέλη αυτή τη χρονιά να μας πούνε σκοπεύουν να τροποποιήσουν ε, την εθνική της νομοθεσία σε σχέση με την άκτα. Σκοπεύουν να επιβάλλουν νέους μηχανισμούς κύρωσης κτλ. πριν ή αφού περάσει άκτα. Τέλος. Ο λόγος που θέλω αυτό το χρόνο είναι ότι θα, υπάρχουν, θα υπάρξουν διαφορές ε, και αλλαγές και θα ήθελα να ξέρω ποιες θα είναι αυτές πριν, πριν να καταλήξουμε στην άκτα. Εντάξει, δεν λέω ότι σήμερα το πρωί θα πάρω απαντήσεις, γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα ε, στο θέμα της άκτα. Αυτό όπως που θέλω να καταδείξω και είναι προς όφελος όλου του σώματος, είτε είσαστε υπέρ είτε κατά, είναι ότι την επόμενη χρονιά ε, να είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνειδητοποιήσει ότι έχει μια ευαίσθητη υπόθεση στα χέρια του για την οποία έχουν δείξει ενδιαφέρον εκατομμύρια πολίτες και έτσι οφείλει να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη θέση που να διέπεται από συνοχή. Το θέμα δεν είναι μόνο να πούμε ναι ή όχι. Αν το ψάξουμε καλά και καταλήξουμε έτσι όπως σας είπα, τότε θα κερδίσουμε σε αξιοπιστία από τους Ευρωπαίους πολίτες και ψηφοφόρους μας. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, εξακολουθεί να μας πιέζει ο χρόνος, θα βάλω το χρονόμετρο και παρακαλώ να αυτοπεριοριστείτε. Αν δεν λειτουργήσει το εθελοντικό σύστημα, θα βάλω εγώ όριο στο χρόνο αγόρευσης. Θα δώσω επίσης προτεραιότητα στους σκιώδεις εισηγητές όταν θα καταρτήσω τον κατάλογο μιλητών. Αρχίζω με τον Κρίστοφε Φιέλεν. ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και ευχαριστούμε, Ντέιβιντ. ομολογώ ότι χαίρομαι που επιτέλους ξεκινούμε με αυτό το θέμα. Το περίμενα τόσο πολύ καιρό, δηλαδή να έχει την ευκαιρία το Κοινοβούλιο να εξετάσει λεπτομερώς αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν διάφορες αξιώσεις, ερωτήσεις, ανησυχίες στο δημόσιο διάλογο που γίνεται και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι δικό μας καθήκον είναι να κάνουμε μια διαλογή, να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Επί τη βάση του κειμένου και της νομικής γνωμοδότησης και όσων έχω ε, καταλάβει μέχρι στιγμής, ε, έχω την εντύπωση ότι τι να πω, 50% είναι μύθοι. Ένας από τους μύθους που άκουσα από την πρώτη μέρα που αρχίσαμε να συζητάμε την άκτα είναι ότι θα αρχίσουν τα τελωνία να ελέγχουν το iPod μου τώρα. Όμως μέσα στο νομικό κείμενο αναφέρεται ρητά ότι τα συμβαλόμενα μέρη δίνανται να ε, προβλέψουν αυτήν την εξαίρεση. Είναι ξεκάθαρο. Άρα καταρρύπτεται ο μύθος. Και ξαναλέω ότι περίπου 50% όλων αυτών των ζητημάτων αξιώσεων και ανησυχιών ε, θα πρέπει να εξεταστούν ε, ε, διεξοδικότερα για να καταρριφθούν οι τυχόν μύθοι. Επίσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη δουλειά μας, να αξιολογήσουμε δηλαδή επακριβώς το περιεχόμενο της συμφωνίας. Και η Επιτροπή και ο Ντέιβιτ μας μίλησαν επί μακρόν για την έλλειψη διαφάνειας και γενικότερα για τη διαφάνεια. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης, πιστεύω. Δείτε στα πρακτικά της προηγούμενη Ολομέλειας, θα δείτε κάποιε παρεμβάσεις, ε, μεταξύ των οποίων και οι δικέ μου, αλλά και κάποιων άλλων, ε, που το κατήγγυλαν αυτό, ότι δηλαδή δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια στο φάκελο άκτα. Ε, ε Ω προ τι εμπορικέ διαπραγματεύσει, νομίζω θα αντλήσουμε από αυτό δίδαγμα και για μελλοντικέ διαπραγματεύσει στο παρελθόν. Τέτοιου είδου διαπραγματεύσει ε, πάντοτε διεξάγονταν κατά αυτόν τον τρόπο. Όμω, από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δημόσια γνώμη άρχισε ουσιαστικά να συμμετέχει στη διαδικασία, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα τώρα. Όμω, οφείλουμε να ομολογήσουμε επίση ε, ότι δεν έχω δει κανένα νομοθέτημα εμπορικού χαρακτήρα να έχει τόση διαφάνει διαφάνεια ήδη έχει η άκτα. Μπορέσαμε, ε, παραδείγματο χάρη, να διατρέξουμε όλα τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η διαπραγμάτευση. Δεν ε, ίσχυε αυτό στο παρελθόν. Πρόκειται για ε, καμπή ρίξει με το παρελθόν, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματευόμαστε τέτοιες συμφωνίες. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Το ΕΛΚ που εκπροσωπώ για αυτό το ζήτημα σαφέστατα θέλει η διεθνή συνεργασία να προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ε, ιδιοκτησίας. Πιστεύουμε δηλαδή στην ε, διεθνή συνεργασία για την προστασία του, το χρειαζόμαστε για την οικονομία καθώς και για την, ε, τους καταναλωτές, όπως είπε ο Ντέιβιντ. Πρέπει να αναρωτιόμαστε αν ε, είναι αυτού του είδου τη διεθνή συνεργασία που θέλουμε για να λειτουργήσει η άκτα, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να βρούμε νέα ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα διανοητικής ε, ιδιοκτησία και πολιτικών ελευθεριών. Δεν χρειάζεται εκ να αναμορφώσουμε την ε, νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μια τέτοια συμφωνία. Πρέπει επίση να θυμόμαστε και να θυμίζουμε και στου πολίτε μα ότι η νομοθεσία τροποποιεί την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Όχι μια εμπορική συμφωνία. Μια νομοθεσία που θα είναι απότοκο ενδεχομένω, αυτή της εμπορική συμφωνία μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή των πολιτών. Προς το παρόν όμω, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να καταθέσει νομοσχέδιο, εκτό βέβαια από την Σουηδία που θέλει να υποβάλει μια μεταρρυθμιστική ε, ε, ε, τροπολογία. Ε, για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει πάντως γενικότερα πρόθεση για να, γίνει, ε, να αναλυφθεί κάποια νομοθετική πρωτοβουλία από επιτροπή ούτε από κανέναν. Αλλά δεν θα σας πιστέψω ε, απαραίτητα και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι να εξετάσουμε σε κάθε λεπτομέρεια την πρόταση. Θα πρέπει να καλέσουμε όλους όσους από την κοινή γνώμη έχουν αξιώσεις, ερωτήσεις, ανησυχίες εδώ, να τους καλέσουμε επίσης να μας διαβάσουν τη θέση τους γραπτός, ούτως ώστε να μπορέσουμε εμείς να εξετάσουμε ε, ε, ενδελεχώς το ζήτημα και ήρθε η σωστή στιγμή να κάνουμε τη διαλογή ανάμεσα σε αυτά που ευσταθούν και αυτά που είναι ανυπόστατα. Πάντως σίγουρα χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία ε, και πρέπει να, απλώς να αποφασίσουμε αν η άκτα είναι η απάντηση. Αν αυτού του είδου τη διεθνή συνεργασία χρειαζόμαστε. Τώρα από πλευρά ε, ECR λέει ο πρόεδρος ο Ρόμπερτ Στέρντι. Πρόεδρε, δεν μπορεί να έρθει ο συνάδελφο, γι' αυτό θα μιλήσω εγώ. Η Επιτροπή είναι θεματοφύλακα ε, των συνθήκων, όπω ξέρουμε, και την ευχαριστούμε που ήθελε ε, να ε, εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσει συνάδουν με τη συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε, Ντέιβιντ, ότι κρύβεται ο διάβολο λεπτομέρειε. Εμά στην άκτα σίγουρα, όχι, δεν έχει αρκετέ λεπτομέρειε. Κατά τα άλλα είναι εύστοχο το σχόλιο σου. Άκουσα τον Ντέβιτ, άκουσα και τον Κρίστοφερ Φιέλνερ, αλλά υπάρχουν και φυσικά όρια για όλες αυτές τις ερωτήσεις που μπορεί κάποιο να θέσει σχετικά με τις μελλοντικέ εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος ε, ίσω να προτίθενται να εισαγάγουν κάποιες προτάσεις, αλλά υπάρχει θέμα ε, συμβατότητα ε, και ευελιξίας για τι μελλοντικέ μα κινήσει. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη, δεν συντρέχει αν θέλετε λόγος για να υιοθετηθεί μία ε, αλλαγή και μην ξεχνάτε με αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τις κινήσεις μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε όπως είπε ο Ντέιβιντ όλες ε, τις καινοτομίες που ανακύπτουν ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον ε, της ευρωπαϊκής καινοτομίας και τεχνολογίας. Πλην όμως θα οφείλουμε να οριοθετήσουμε τη διαδικασία γιατί είναι μεταβαλλόμενο και το πεδίο στο οποίο σημειώνονται αυτές οι εξελίξεις. Ε, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ πάντως ε, με την ε, δίκαιη νομίζω και ακριβή περιγραφή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κατάστασης και όλες αυτές οι αποφάσεις των οποίων θα επιληφθεί το δικαστήριο. Μας βρίσκουν σύμφωνες οι ιδέες σας. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα, πόσο γρήγορα θα περάσει αυτό από εσά. Και ε, οι προθεσμίες για τη μετάφραση ε, που είπατε που μας δώσατε χθε ε, είναι ενδιαφέρουσες και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επισταμένα να ασχοληθεί με το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Γιάννη Ξαντώ από τους επράσινους Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα σας εξυπηρετήσω. Ξέρετε, θα μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα, λιγότερο από όσο περιμένετε, απλώς ένα διαδικαστικό και ρωτώ τον Επίτροπο. Ε, στο άρθρο 118 της Συνθήκης αναφέρεται, Ρίτα, ότι σε κάθε φάση διαπραγμάτευσης οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας οφείλεται να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για τις αναληφθήσεις πρωτοβουλίες. Την συμφωνία πλαίσιο που είναι δεσμευτική για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αναφέρεται ρητά στο παράγραφο 13 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ε, απόφαση προτού ενημερώσει το Κοινοβούλιο γραπτός. γραπτός. Εσείς αναλάβατε την πρωτοβουλία που το, σας το ζητούσαμε εξάλλου ε, εδώ και ένα χρόνο για να επιληφθεί το ζητήματο στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε υπέρα. αλλά γιατί να το, το μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ, ε, από τον τύπο, γιατί δεν γνωρίζουμε γνωρίζουμε ποια, ε, ποιο είναι το νομικό αίτιο για την προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι παραβιάζεται τρόπον ε, την την ε, συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο περί διαβουλεύσεως. Εφόσον έχει κινηθεί η διαδικασία, θεωρώ ότι αντιβαίνει αυτή η κίνηση στην αίσια λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Θα περιοριστώ σε αυτό και επί τη ουσίας θα μιλήσει ο συνάδελφος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Ντεγκούχτ με ενημέρωσε πριν ανακοινώσει την πρωτοβουλία εμένα. Ο Κάρις Λίτερ τώρα. Λοιπόν, Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι η συμφωνία αυτή είναι σαφής, γιατί κάθε φορά που μιλάω με ένα νέο δικηγόρο, ερμηνεύει την συμφωνία με διαφορετικό τρόπο. Εγώ βέβαια δεν είμαι δικηγόρος, αλλά δεν ξέρω, εσείς είστε δικηγόρος, άρα φαντάζομαι ότι έχετε τη δική σα ερμηνεία και άλλοι έχουν τη δική τους. Ακόμα και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου λέει, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σαφείς ε, αποδείξεις ότι παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και προσθέτουν βέβαια ότι υπάρχουν ε, αρκετά σημεία ε, που χρήζουν ερμηνεία και τελικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίσει για τη σωστή ερμηνεία. Και υπάρχουν κάποιες αρχικές εκδοχές αυτής της συμφωνίας που είναι διαφορετικές από αυτή που έχουμε τώρα. Άρα δηλαδή σας το λέω για να δείτε ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ε, η ορισμός των ε, έμεσων ε, κερδών ή των κατασχεθέντων προϊόντων δεν είναι σαφές. Και επίσης, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν επηρεάζονται με μονομένοι ταξιδιώτες, τότε γιατί δεν χρησιμοποιούμε στα αγγλικά το ΣΑΛ. Είναι πολύ καλύτερο στο ΣΑΛ, ε, είναι πολύ πιο ασφαλές για μας. Κατόπιν, η συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Αυτό είναι κάτι το πολύ πιο ανοιχτό από το να περνάει κανείς ε, από τα δικαστήρια όπως είπατε και αλλά η ΑΚΤΑ διαφέρει από την ε, οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης ε, ενδέχεται να υπάρξει και περιορισμός πρόσβασης στην ενημέρωση και τα Ηνωμένα Έθνη ανησύχησαν γι' αυτό, διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε εμπορικές συμφωνίες που θα περιορίσουν τη δυνατότητα των τελικών χρηστών ε, να αποκτήσουν πληροφορίες. Γι' αυτό λοιπόν Ίσως ε, πρόκειται για μια εσωτερική συμφωνία η οποία θα περιορίσει την πρόσβαση στην ενημέρωση κυρίως για τους ε, τελικούς χρήστες. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, χέγγια επ' αυτού. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους τεχνικούς φραγμούς για την διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων. Αυτό θα επηρεάσει την καινοτομία. Γιατί αν τελικά ο στόχο τη ΑΚΤΑ είναι να ενθαρρύνει την καινοτομία, εγώ βλέπω ότι θα περιοριστεί η καινοτομία, γιατί σα λέω ότι θα υπάρξει παράπλευρη χρήση προγραμμάτων που θα παραβιάσουν τα ψηφιακά δικαιώματα που ενδεχομένως αυτό να μην ήταν ο πρωταρχικός στόχος αλλά θα προκύψει. Έχουμε ένα πρόσφατο πρόγραμμα το οποίο ε, δεν, ε, για αυτούς τους λόγους δεν είναι δυνατόν να κατέβει στα iPhone. Αν λοιπόν θέλουμε να προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, αυτή η συμφωνία δεν προσφέρει τέτοια δυνατότητα. Γιατί, παραδείγματο χάνει στη δική μου τη χώρα και ίσω και σε άλλε, βλέπουμε ότι οι χώρες αυτές ε, και αναφέρθηκε προσωπούν το 50% του διεθνού εμπορίου. Όμως, μόνο το 5% παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων εμπίπτουν και κατασκευάζονται σε αυτές τις ε, χώρες Το 50% δηλαδή τα περισσότερα κατασκευάζονται σε άλλες χώρες που δεν έχουν ε, υπογράψει τη συμφωνία Άκτα. Άρα δηλαδή, αν ο στόχος είναι να διαδώσουμε την άκτα χρησιμοποιώντας ε, διμερείς συμβάσεις, νομίζω ότι αυτό ε, δεν είναι δημοκρατικό όπως προσπαθούμε να το κάνουμε. Να το πω αλλιώ. προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τις διατάξεις ε, της ΑΚΤΑ και να τις ε, προσθέσετε σε διμερείς συμφωνίες. Αν το σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, είναι πολύ αντιδημοκρατικό για να αλλάξετε την νομοθεσία άλλων κρατών. Γι' αυτό σας ερωτώ. Επίσης ανησυχώ, διότι ενδέχεται να μας δεσμεύσουν διατάξεις που τώρα είναι υπό αναθεώρηση. Βεβαίω ε, έχουμε κάποιε καλέ ρήτρε ασφαλεία ε, στην ηλεκτρονική εμπορία, αλλά τι θα γίνει αν αυτέ ε, επηρεαστούν από την άκτα. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να δεσμευτούμε περαιτέρω όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία της ενημέρωσης. Πρόεδρος, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Καντάρα Αρίφ, ε, γιατί βρίσκεται υπό πίεση χρόνου και διότι παλαιότερα ήταν και εισηγητή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από μερικές εβδομάδες αποφάσισα να εκφράσω την άποψη ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το καρναβάλι της απόφασης αυτής. Και σήμερα δεν μπορώ να πω ότι νιώθω ευτυχής, αλλά βλέπω μια εξέλιξη σε αυτά που λένε διάφοροι συνάδελφοι εδώ, οι οποίοι μας είχαν επιβάλει ένα χρονοδιάγραμμα, το ΕΛΚ δηλαδή, να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, η Κομισιόν. Οπότε εδώ ευχαριστώ τον κύριο Φέλνερ που εξέφρασε και αυτός τις αμφιβολίες του. Χαίρομαι επίσης και για την εξέλιξη που βλέπω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να υποβάλει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να υπάρξουν, όπως θα κάνουμε και εμείς, για να υπάρξουν διευκρινήσεις στο νομικό επίπεδο. Εννοείται ότι έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες όσον αφορά την ε, ατομική ελευθερία, ε, το δικαίωμα, το συμβατό με συμφωνίες όπως είναι η τρίψη, η γεωγραφική διάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Τους ένα σωρό αμφιβολίες και αμφισβητήσεις που εγείρουν οι πολίτες. Παρ' όλα αυτά είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Βέβαια ο επίτροπο λέει ότι δεν θα αλλάξει και τίποτα. Λοιπόν, όταν μα υποβάλλεται ένα κείμενο το οποίο κρίνεται επικίνδυνο ή τέλο πάντων γύρει ανησυχίε και αμφισβητήσει, ε, αλλά που η Επιτροπή μα λέει μα δεν θα αλλάξει και τίποτα, ε, α τον καταλήψουμε τότε. Γιατί να το έχουμε. Το θέμα είναι να βελτιωθεί η κατάσταση. Πάντως, χαίρομαι σήμερα γιατί έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Εδώ υπάρχουν εξελίξεις. Το ότι σήμερα γίνεται δημόσια συζήτηση και με περισσότερη διαφάνεια, αυτό είναι πιο θετικό από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε. Ε, το αποφασίσαμε στους συντονιστές και το ΕΛΚ ε, εφόσον δεν τον αποφάσισε. Ας Προχωρήσουμε τώρα στον κατάλογο. Γιώργος Λάις; Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να βάλω ε, περιορισμό χρόνο από τώρα και στο εφεξής λέει πρόεδρος. Λοιπόν, ε, ο Λάχτριτ, εγώ παρακολούθησα τη συζήτηση και πραγματικά εξεπλάγει, γιατί εδώ συζητάμε πολύ συμπαθητικά, χαλαρά, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι ακριβώς το αντίθετο. Εντάξει, και εγώ και χαλαρός είμαι, αλλά ξέρετε, ε, δεν θέλω να γίνεται έτσι η συζήτηση. Κοίταξα τη συμφωνία άκτα και εγώ νομικός, νομομαθής είμαι και εδώ ξέρετε πριν την πρόκειται να σας πω, μας παρασύρουν. Η Ευρώπη παρασύρθηκε να καταλήξει σε μια συμφωνία που αφορά υποτίθεται τα προϊόντα μας, την προστασία των προϊόντων μας και τελικά τι προέκυψε. Προστατεύονται καλύτερα οι φαρμακευτικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, στην Ασία και αν στο μέλλον ας πούμε, η Lady Gaga και ο κύριος ε, ε, Spielberg έχουν πρόβλημα, ξέρετε ποιο θα είναι το πρόβλημα τους αν θα αγοράσουν 8 αεροπλάνα ή 15. Γιατί να σας πω το εξή. Ποιο πιστεύει ότι με αυτή τη συμφωνία θα παίξει ρόλο η προστασία των προϊόντων μας. Μα με συγχωρείτε, η Ελβετία δεν παραποιούν ευρωπαϊκά προϊόντα. Ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε το κάνουν αυτό. Ξέρετε ποιοι το κάνουν. Το κάνουν αυτοί που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία και ε, που προφανώς τη συμφωνία αυτή θα την προσβάλλουν και στον ΠΟΕ. Και αυτό δεν το συζητήσαμε ακόμα και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Ε, τότε τι, τι θέλουμε αυτή τη συμφωνία. σα το λέω ξεκάθαρα. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις, αλλά εγώ είμαι κατά μία ε, συμφωνίας η οποία ξαφνικά τα αστικά δικαιώματα τα μετατρέπει σε ποινικά διώξιμα απλά και μόνο για να προστατευτούν οι ολίγοι. Και εγώ είμαι κατά μια συμφωνία η οποία εξαναγκάζει ιδιωτικέ επιχειρήσεις ε, ε, στο μέλλον να κάνουν κατασκοπία για άλλους ιδιώτες για το κράτος. Και στην Αυστρία χρησιμοποιούμε μάλιστα και μια έκφραση την έκφραση του δοσίλογου. και αυτή την εποχή δεν θέλω να την ξαναφέρνω στο μυαλό μου. Ε, μην ξεχνάτε όμως ότι αυτή είναι μια συμφωνία του 20ου αιώνα η οποία πλέον δεν σέβεται τον 21ο αιώνα. Σήμερα οι νέοι ε, χειρίζονται το διαδίκτυο τελείως διαφορετικά. Και γι' αυτό δεν είναι πλέον επίκαιρη η συμφωνία. Νομίζω λοιπόν ότι νομικά καθαρά δεν θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε τις απαγορεύσεις και να το κάναμε αυτό νομίζω ότι δεν θα ήταν στο ύψος της ε, ε, στάσης ζωής ε, των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, θα προσπαθήσω να τηρήσω τα τρία λεπτά και αν μακρηγορήσω λιγάκι ε, παρακαλώ να δείξετε υπομονή. Γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο στην Ευρώπη συζητιέται ε, με μεγάλη φόρτιση. Η δική μας ε, η Επιτροπή δεν ασχολήθηκε μέχρι σήμερα με θέματα δικαιωμάτων του πολίτη. Και υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά σε αυτή την, ε, συμφωνία. Και αυτές οι επιφυλάξεις έχουν σχέση με τις ευρείες ελευθερίες του πολίτη. Πρέπει να το στήσουμε αυτό. Εχθές για το Περού και την Κολομβία μιλάγαμε δυόμιση ώρες. Νομίζω, σας παρακαλώ, να προβλέψουμε τουλάχιστον τον ίδιο χρόνο για τη συμφωνία ΑΚΤΑ. Πάω τώρα στην ουσία του θέματος. Κύριε Επίτροπε, εχθές σας άκουσα πολύ προσεκτικά και θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ανάμεσα στους υπέρμαχους και τους πολέμιους της ΑΚΤΑ δεν αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Στην Ευρώπη όλοι τάσσονται υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. Μα είναι αυτονόητο. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα έχει σχέση ή αφορά εκείνους που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα στις ε, ε, νομικές διατάξεις ε, που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Αυτοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνει καμία προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα που έχει προκύψει με το διαδίκτυο. Πιστεύουν ότι θα πρέπει να προστατευτούν καλύτερα τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτή είναι η μεν. Και οι δε πιστεύουν ότι θα πρέπει καταρχήν να εξεταστεί ποιες διατάξεις ισχύουν αυτή τη στιγμή και να αναλυθεί, να βολιδοσκοπηθεί ποιες είναι οι αλλαγές ε, που προέκυψαν λόγω του διαδικτύου. Ή δε θέλουν, το σκεφτούν πολύ συνετά τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα και μόνο αφού γίνει αυτή η ενδελεχής έρευνα για τις ε, νομικές διατάξεις, μόνο τότε θα σκεφτούν ή θέλουν να σκεφτούν ενδεχομένως να ε, θεσπιστούν νέες διατάξεις. Και όσον αφορά τα εμπορικά σήματα. Και εκεί υπάρχουν διαφωνίες, αλλά κατά κύριο λόγο πρόκειται για την ελευθερία στο διαδίκτυο. Εγώ λοιπόν συμφωνώ με τον Επίτροπο που λέει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ε, τον οποίο επικαλούνται οι πολέμοι είναι ότι η Συμφωνία Άκτα δεν ε, ισχύει, αγνοείται διότι ότι ε, κατ' ουσίαν αμφισβητούνται τα ε, δικαιώματα του πολίτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η συμφωνία άκτα είναι καλή, είναι κακή, διότι είναι ασαφής, διότι έχει πάρα πολλές ασάφειες. Παραδείγματο χάρη, το ύψος των αποζημιώσεων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Επίσης, ε, τίθεται το ερώτημα ε, ποιες είναι οι νομικές αλλαγές που θα προκύψουν. Ε, εξετάζεται το κατά πόσο ενδεχόμενο σε περιπτώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων να μπορεί κανείς να καταφύγει στα δικαστήρια. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυνατότητες τις οποίες εξετάζει ο θεματοφύλακας των της προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη. Για τη τελική ανάλυση πρόκειται και γι' αυτό, για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κυκλοφορούν πάρα πολλές εφήμες για αυτή τη συμφωνία πολλά από αυτά που λέγονται είναι γνωστά και σε τελική ανάλυση πρέπει να έχουμε κατά νου ποιες ήταν οι προθέσεις εκείνων που πρώτο εμφάνισαν αυτή τη συμφωνία. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε που μακρηγορώ, αλλά το θέμα αυτό συζητιέται με πάθος ε, στην ε, Πολωνία και πρέπει να τα πω. Πρόεδρε, ναι, αλλά θέλουν και άλλα να μιλήσουν. Ναι κύριε Πρόεδρε, αλλά επιτρέψτε μου τουλάχιστον να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ολοκληρώνω λοιπόν. Η συμφωνία Άκτα είναι μια συμφωνία που αν δει κανεί τις προθέσεις των κρατών που ξεκίνησαν τη συμφωνία αυτή, η συμφωνία παραβιάζει σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα ε, που έχουν κατοχυρωθεί σε σχέση με το διαδίκτυο. Ο δρόμος είναι πολύ σημαντικός, ε, μάλλον ο σκοπός, αλλά και ε, το, τα μέσα που οδηγούν στο σκοπό. Η συμφωνία άκτα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον τρόπο με τον οποίο το επιθυμούν οι πολίτες. Έχουμε τώρα αντιδράσεις ε, σε διάφορες χώρες. Ε, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και της Πολωνίας. Η Πολωνία δεν επικύρωσε τη συμφωνία αυτή και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή τη συμφωνία πρέπει να τη θεωρούμε παρελθόν. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, ένταση που υπάρχει ανάμεσα στην προστασία, ε, την ελευθερία στο διαδίκτυο και την προστασία των ε, ατομικών δεδομένων. Να δούμε λιγάκι τι σημαίνει ιδιωτική χρήση. Και όταν θα έχουν αναλυθεί όλα αυτά, τότε θα πρέπει πάνω σε μια νέα σταθερή βάση να επεξεργαστούμε μια νέα συμφωνία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, εντάξει, αλλά έτσι όπως κάνετε, ε, ουσιαστικά οι υπόλοιποι θα πρέπει να μιλήσουν λιγότερο. Είναι άδικο για τους άλλους. Θα έχουμε την ευκαιρία ξανά και ξανά να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα ίσης μεταχείρισης και δικαιοσύνης απέναντι στους άλλους. Σάιμον Βουσάτιλ από την ΛΥΜΠΕ. Δεν είσαστε μέλος επιτροπής αυτής, αλλά καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όντως είμαι ο συντονιστής του ΕΛΚΑ στην ε, Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη. Και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα που συζητάμε. Όταν για πρώτη φορά διάβασα τη συμφωνία αυτή, σκέφτηκα γιατί να είμαι κατά. Εδώ θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παραποίηση, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, οπότε γιατί να είμαι εναντίον. Μετά όμως υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην ε, δημόσια συζήτηση που έγινε και επικεντρώνομαι στο θέμα των ελευθεριών ακριβώς του πολίτη που περιλαμβάνονται στη συμφωνία αυτή και την ελευθερία στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η Επιτροπή πρέπει να καταλάβει ότι η ελευθερία στο διαδίκτυο δεν ε, Οπότε φοβάμαι ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή, ακόμα και αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την πειρατεία και την παραποίηση προϊόντων. Αυτό είναι το πρώτο. Από πλευρά δηλαδή ελευθεριών του πολίτη, η συμφωνία αυτή εγείρει ανησυχίε. και οι ανησυχίες αυτές πρέπει να καθησυχαστούν. Δυστυχώ παρά την πολύ ενδιαφέρουσα χθε παρουσίαση που έκανε ο Επίτροπος, δεν βλέπω να έχουν καθισχαστεί οι ανησυχίες μας. Δυστυχώς, η δημόσια συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και δυστυχώς έχει δηλητηριαστεί. Και θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση. Θα έπρεπε να διορθώσουμε τα... οι στραβές αλήθειες που κυκλοφορούν και έπειτα με το που ξεκινάει κανεί, αμέσω του επιτίθενται. Δηλαδή δεν καταφέρουμε να την κάνουμε καλά αυτή τη συζήτηση και υπάρχει και κακή ε, επικοινωνία, ανακοινώσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει την στρατηγική τη επικοινωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Γιατί αλλιώ όντω μπορούμε να τη θεωρήσουμε ξεχασμένη αυτή τη συμφωνία. Κοιτάξτε κύριε Επίτροπε, αν είσαι μέσα σε ένα χώρο όπου όλοι ουρλιάζουν, όσο λογικά πράγματα κι αν λες, δεν θα σε ακούσει κανείς. Και φοβάμαι ότι αυτό ακριβώ συμβαίνει και με τη συμφωνία αυτή άκτα. Πρόεδρος, κατάλογος ομιλητών έχει κλείσει. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στο ΕΛΚΑ, την κυρία Νεσφέρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, σας άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον χθες όταν κάνατε την ομιλία σας. Εκτίμησα την ενημέρωση που μας προσφέρατε και εκθέσατε την άποψη που θέλησα να ε, υπερασπιστώ και εγώ στην ε, Λετωνία, τη χώρα μου. Δεν είναι πεπισμένοι οι άνθρωποι για ποιο λόγο χρειαζόμαστε αυτή την πρόταση. Ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα, μια τόσο σημαντική συμφωνία θα έπρεπε ε, να έχει εξηγηθεί διεξοδικά στο κοινό. Έπρεπε να το είχατε προβλέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα γινόταν έντονος δημόσιος διάλογος και θα υπήρχε ισχυρό ενδιαφέρον από πλευρά κοινή γνώμη. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Επειδή εσείς ασχολείστε με την επικοινωνία με το κοινό, θα σας έλεγα λοιπόν ότι δεν κατανοούν όλες τις διαστάσεις του ζητήματος οι πολίτες. Υπάρχουν δύο ε, ειδών ε, προβλήματα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχει γενικό πρόβλημα γιατί δεν έχει διαβάσει τη συμφωνία και δεν κατέχει καθόλου το αντικείμενο. Μια δεύτερη κατηγορία είναι φιέστατοι άνθρωποι που έχουν ήδη διαβάσει τη συμφωνία άκτα που κατέχουν το αντικείμενο και που ισχυρίζονται ότι είναι εξαιρετικά Σαφέ ε, το κείμενο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι παραβιάζονται οι πολιτικές ελευθερίες. Άλλοι πάλι ε, αναρωτιούνται τι σημαίνει αυτός ο ορισμός περί παραποίηση counterfeiting. Ε, υπάρχει μεγάλο περιθώριο παρερμηνία τη έννοια. Κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν τρίτα μέρη, τρίτες χώρες ενδεχομένως που θέλουν να προστατεύσουν να προστατευτούν μάλλον από τον ανταγωνισμό. Και σας παραπέμπω στο άρθρο 12, υποσημεία 1, 2 και 3. Εκεί αναφέρεται ότι προβλέπεται άμεση αναστολή του άκτα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ποινικοποίηση αλλά όμως δεν αναφέρεται η αναστολή δραστηριότητας ε, ε, πόσο θα διαρκέσει. Όταν μιλάμε για commercial scale, εμπορική κλίμακα, τι εννοούμε ακριβώς μέσα στο κείμενο. Επίσης, ε, είναι αληθεύει ότι κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα να εγκαταστήσουν φίλτρα, παραδείγματο χάρη, για να ελέγχουν τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Ε, δεν ξέρω αν ερμηνεύω σωστά αυτά τα πρότυπα, ούτε αν τα ερμηνεύουν σωστά οι επαγγελματίε. Έχουν δίκιο οι επαγγελματίε ότι θα ε, εισαχθούν τέτοια μέτρα και ότι θα περιοριστούν οι ελευθερίε ε, στο διαδίκτυο. Υπολείπεται μεγάλο έργο σε κάθε περίπτωση, ε, αλλά φοβούμε ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Το, το νομοθέτημα λοιπόν κατά της παραποίησης σίγουρα είναι εκ των νόνου κάνευ. Απλώς ελπίζω ότι θα καταφέρουμε ε, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκαίρω. Δεν έγινε εγκαίρω η διαβούλευση με το κοινό και για κάποιου δημαγωγικού ε, λόγου ε, δεν δίνονται επαρκεί εξηγήσει στο κοινό για να μπορέσει να τοποθετηθεί στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα είμαι σύντομη γιατί με πρόλαβαν οι προλαλήσαντε. Θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει. Πρώτον, έχουμε ακούσει πολλές τοποθετήσεις ε, από πολίτες ε, και ε, εμπλεκόμενοι φορείς, επιχειρήσεις παραδείγματο χάρη λένε ότι η άκτα είναι τέλεια λύση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μήπως η άκτα έχει γίνει σαν χριστουγεννιάτικο δέντρα όπως λέμε ή προσπαθούμε με ένα σμπάρο να πιάσουμε δύο τριγώνια όπως λέμε στα ελληνικά. Προσπαθούμε δηλαδή να καλύψουμε τα πάντα με το άκτα αγνώντας τις παράπλευρες απώλειες που επισύρει. Ε, θεωρείτε εσεί ότι θα είναι μια θεσπέσια λύση η άκτα για όλε τι ανησυχίε που έχουν αναφερθεί για τα παραποιημένα παραδείγματο χάρη φάρμακα που κυκλοφορούν ε, στο εμπόριο. Άλλη ερώτηση τώρα. Είναι δυνατόν ε, ε στο όνομα μιας συμφωνίας κατά της παραπίεση ε, να μεγενθύνεται διαρκώς η πειρατεία και Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα η ΑΚΤΑ, οι συμπράξει δε δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η εποπτεία της διαδικτυακή συμπεριφορά πολιτών και επιχειρήσεων ε, προστατεύεται. Οι πάροχοι υπηρεσιών σίγουρα δεν θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν τη βρώμικη δουλειά που κανονικά είναι καθήκον του κράτου. Υπάρχει διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και δεν θέλουμε ε, ιδιωτικοί φορεί να αναλάβουν θεσμικό ρόλο παρακολουθώντας τη διαδικτυακή συμπεριφορά των ε, ανθρώπων. Ε, από το ΕΛΚ τώρα σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ συμφωνώ με πολλά από τα θέματα που ετέθησαν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα έτσι ώστε να καταλήξουμε στη λήψη απόφασης. Επίσης ε, γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πάρα πολλές ε, θεωρίες ε, συνωμοσία μεταξύ αυτών και το ότι πίσω από όλα αυτά υποτίθεται κρύβεται ή κρυβόταν κατά το παρελθόν ένα πολύ ισχυρό λόμπι, το οποίο ε, επηρέασε τη σύνταξη των κειμένων και σε διάφορα άρθρα αναφέρεται συνεχώς το όνομα μιας συνεργάτη δόσας η οποία για πάρα πολλά χρόνια ε, δραστηριοποιείται ε, ως δικηγόρος ε, πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρου τη μουσική βιομηχανία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ τίθενται διάφορα ερωτήματα και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσει η Κομισιόν απαντήσεις. δηλαδή, ε, κατά πόσον πράγματι υπήρξε ανάμειξη άλλων. Και κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και σε σχέση με την ΑΚΤΑ ε, είναι ότι τα GIs, ε, οι, οι ονομασίες γεωγραφικής προέλευσης ε, στο γεωργικό τομέα, αυτά θα επηρεαστούν, αυτές οι ονομασίες. θα υπάρξει δηλαδή παρακολούθηση και κάποιο είδους αντιστάθμιση. Τελευταίος ομιλητής ε, εκ μέρους της Ενωμένης Αριστεράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Νομίζω, κοιτάξτε, ε, όποιος ε, σπήρει ανέμου θα εθερίζει θύελες. Δεν πρέπει λοιπόν να εκπλησώμεθα για το ότι το θέμα αυτό έχει προκαλέσει ένταση. Και δεν είναι κακό. Θεωρώ ότι αν θέλουμε οι πολίτες να ε, δείξουν κατανόηση, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Και το δεύτερο, κάτι που με απασχολεί, κυρίως ε, σε σχέση με την πειρατεία προϊόντων. Οι χώρες οι οποίες κατ' ουσίαν θίγονται εξαιρούνται και η προσέγγιση αυτής της συμφωνίας ΑΚΤΑ τελικά και αυτή είναι μάλλον αδιάφοροι. Γιατί, διότι όταν τον Οκτώβρη, ήδη τον Οκτώβριο του 2010, ο Υπουργός Εξωτερικών της ε, Βραζιλίας ε, ανέφερε ότι η συμφωνία αυτή αφορά τα δικαιώματα ανάμεσα στους δικαιούχους ε, και τους τρίτους που ασχολούνται με την προσέγγιση των προϊόντων ή η Κίνα, η Ινδία. Αυτοί αναφέρουν ότι αυτή από την συμφωνία τη συμφωνία απλά την ε, λαμβάνουν υπόψη. Αλλά δεν είναι το να λαμβάνουν υπόψη. Αυτοί, αυτές οι χώρες κατηγορούνται για πειρατεία. Άρα δηλαδή αυτές οι χώρες ε, καλούνται να ε, θεσπίσουν νέους κανόνες. Και κάτι άλλο. Ε, οφείλουν να επηρεάσουν και τους πολίτες των χωρών τους. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Εχθές, μιλώντας ε, για το ε, παγκόσμιο εμπορικό σύστημα του Πασκάλα Μη, ναι, προφανώς η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις αυτή λοιπόν η προσέγγιση της ΑΚΤΑ δεν είναι σωστή. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, υφιστάμενες ε, δομές ε, έτσι ώστε να επιτύχουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Και φτάνουμε λοιπόν στο κατά πόσον η συμφωνία ΑΚΤΑ είναι συμβατή με τη συμφωνία TRIPS. Και σας λέω ότι υπάρχουν διαφορές, ε, υπάρχει διαφορές το 8-1, 8-2, 8-11, το 12-1. Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία για ε, τα θέματα που αφορούν και η άκτα και οι τρίψ. Δεν έχω τώρα χρόνο για να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι ο Ευρωπαίος ε, εντεταλμένος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Αυτά που λέει για την μουσική βιομηχανία προβάλλονται περισσότερο από τα δικαιώματα των πολιτών. Δίκαιο έχει ο Προελίσσα που λέει ότι πράγματι χρειαζόμαστε κοινή πρωτοβουλία για την ε, δημιουργία ενός σύγχρονου δικαίου περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Να είναι προσαρμοσμένο στον 21ο αιώνα, στο διαδίκτυο και όχι να εξακολουθούμε να διαφυλάσσουμε το status quo, το ε, ξεπερασμένο. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω και εγώ τις εργασίες ε, για τη Συμφωνία Άκτα και με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω σήμερα το απόγευμα την ομάδα εργασίας όπου φαντάζομαι ότι θα ενημερωθούμε για νέα δεδομένα. Ευχαριστώ, Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να έχουμε την ευκαιρία επί της ουσίας να συζητήσουμε το περιεχόμενο της Συμφωνίας Άκτα. Η συζήτηση αυτή ε, φυσικά και έρχεται κάπως αργά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στις μέλη, ιδιαίτερα σε αυτές που δεσμεύτηκαν με την υπογραφή του στο Στόκιο, η συζήτηση αυτή είχε ήδη γίνει. Συμφωνώ πάντως με τον κύριο Ζελεύσκη για το ότι ως επιτοπλίστων στις χώρες αυτές υπάρχει πολιτική συνένεση. Η χώρα μου, η Βουλγαρία και η Πολωνία, για παράδειγμα. Η πολιτική αυτή συνένεση έχει να κάνει με το γεγονός ότι λάβαμε υπόψη μας τις ανησυχίες που γύρονται για τη συμφωνία αυτή. Ακούσαμε τις διαμαρτυρίες των πολιτών οι οποίες ανάγκασαν την κυβέρνηση να παραιτηθεί από τις αρχικές της ε, προθέσεις να επικυρώσει τη συμφωνία αυτή. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ισορροπία στη συμφωνία αυτή ανάμεσα στους θεμητούς στόχους που είναι η προστασία ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας από την αλλά από την άλλη μεριά κάτι που ίσως είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι το σημαντικό δικαίωμα ενημέρωσης, ελευθερίας έκφρασης. Με μια τέτοια διεθνή συμφωνία παραβιάζουμε όμως τη δεύτερη ελευθερία. Τίθεται εν κινδύνο. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό. Στη συμφωνία αυτή Έχουμε διατυπώσεις ε, και φράσεις ε, ασαφείς. Όταν λέει ότι κάτι ίσως συμβεί κάτι μπορεί να συμβεί, ε, μετά όλα αυτά επιδέχονται ερμηνεία. Και η ερμηνεία αυτή θα είναι διαφορετική. Κάποιοι θα θελήσουν να δώσουν κατασταλτικό χαρακτήρα στις ε, διατυπώσεις αυτές. Δεν θα πρέπει οι πολίτες να φοβούνται, όπως συμβαίνει τώρα, επειδή δεν ξέρουν πώς θα ερμηνευτεί η συμφωνία αυτή και πώς θα την εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα όταν ακόμη τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις και τους ε, παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο να εκφράζουν φόβους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άργησε να έρθει και να μας ε, ζητήσει να συζητήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωβουλευτές πρέπει να έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά για πολλά θέματα να ε, μπορούμε ε, έγκαιρα να ξεκινάμε τη συζήτηση και να μας δοθεί ευκαιρία και τώρα να ακούσουμε και να ξανακούσουμε τον Επίτροπο για να μας διαβεβαιώσει ότι οι ανησυχίες μας αυτές λαμβάνονται υπόψη και καθισχάζονται. Φυσικά και συγχρόνως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφανθεί και θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε στην τελική μας θέση αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι το δικαίωμα των ανθρώπων. Αυτό θα καθοδηγήσει την απόφασή μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Φλίγκερ. Κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχω δύο ε, ερωτήσεις ουσίας που με απασχολούν. Η μία είναι η εξής. αν μετά το άρθρο 26, μάλλον αν σταματούσε η συμφωνία στο άρθρο 26 δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Εκεί που γινόταν λόγος για την ε, ε, παραποίηση προϊόντων. Αλλά αυτή την παραποίηση την μεταφέρατε ε, στον ψηφιακό τομέα. Και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Γίνεται κάτι τέτοιο ή μήπω πρέπει κανείς να αναζητήσει μια νέα προστασία νομική προστασία που να έχει σχέση με τα ψηφιακά δικαιώματα. Γιατί πλέον ε, δεν είναι άμεση αυτή η σχέση ανάμεσα στον προσφέροντα και τον χρήστη. Το ίδιο πρόβλημα είναι και με τα φωτοαντίγραφα. Ε, γι' αυτό στη Γερμανία, παρήματος χάρη, τα μηχανήματα που κάνουν φωτοαντίγραφα είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν εισφορές για να πηγαίνουν εισφορές αυτές στους ε, δικαιούχους ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Και ξέρω κύριε Επίτροπε ότι και εσείς ε, σκεφτόσατε λιγάκι το θέμα των δικαιωμάτων του δημιουργού σε σχέση με το διαδίκτυο. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον είναι σωστό να μεταφέρει κανείς ένα απαρχαιωμένο σύστημα σε μια νέα κατάσταση. Ξέρουμε ότι το θέμα ε, των δικαιωμάτων στο δίκτυο, έτσι κι συζητείται Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή ε, καταβάλουμε τεράστιες ε, προσπάθειες, κάνουμε πυρουέτες, τεράστια η προσπάθεια, προσπάθεια που είναι συνδεδεμένη και με ασαφείς προθέσεις. Μα αξίζει όλο αυτόν τον κόπο αν δεί κανεί στην υπεραξία που προκύπτει. Γιατί στη τελική ανάλυση μόνο λίγες χώρες ενδιαφέρονται και εκείνες οι οποίες κατ' ουσίαν προκαλούν τα προβλήματα αυτές εξαιρούνται ή δεν συμμετέχουν. Μα σε τελική ανάλυση μήπως ε, πρόκειται μόνο για μια πολιτική φύσεως κίνηση που ε, χαρακτηρίζει τους καλούς και τους κακούς και στη τελική ανάλυση βοηθάει αυτό. Αυτές οι δύο ερωτήσεις ουσίας, ε, κύριε Επιτρόπη, με απασχολούν πάρα πολύ. Ο κύριος Κασπάρη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο, τους κυρίους Μάρτιν Φέλνερ, Μπουζιτήλ και Λάγκε. Ε, πράγματι, τους, ε, τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε για να εξετάσουμε σε βάθος την άκτα. Γιατί από τη μια υπάρχουν, ε, υπάρχει κίνδυνος ε, για τις θέσεις εργασίας ε, και οποτεδήποτε αναφέρεται ότι δεν συμμετέχουν οι παραγωγοί των παραποιημένων προϊόντων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριοι ε, και στο θέμα της ε, προστασίας του κλίματος οι κύριοι γιατί και αυτοί δεν συμμετέχουν ούτε οι Κινέζοι ούτε οι Αμερικανοί. Αλλά εμεί συνεχίζουμε. Ε, γι' αυτό λοιπόν αυτό το επιχείρημα, σα παρακαλώ πολύ, δεν ισχύει να το ξανασκεφτείτε. Και κάτι άλλο, το θέμα τη ελευθερία στο διαδίκτυο. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο κύριο Μπουζουτήλ. Δηλαδή για μα, για το ΕΛΚ, του τελευταίου μήνε, ε, τα τελευταία χρόνια, έχει προκύψει με απόλυτη σαφήνεια ότι πρέπει να προκύψουν ε, περισμοί και αν γίνει βέβαια κάτι τέτοιο, ενδεχομένω να απορριφθεί η συμφωνία. Αλλά πρέπει να την εξετάσουμε. Και κάτι άλλο. Σήμερα, από σήμερα, από την 1η Μαρτίου του 2012, ισχύουν νέε διατάξει χρήση του Google και ε, όλοι οι πολίτες ε, από ό,τι φαίνεται εμπιστεύονται περισσότερο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και την Κομισιόν. Αυτό με απασχολεί. Για δέστε τι κάνει από σήμερα η Google. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αλλά από σήμερα η Google το κάνει ε, πιο διεισδυτικά και με ανησυχεί αυτό. Η Google μπορεί να κατασκοπεύει τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία για να μας ε, προσφέρει, να μας ε, προσφέρει καλύτερες ε, προσφορέ στην ΠΕΝ. Αυτό μπορεί να αρέσει σε μερικούς, αλλά με συγχωρείτε κυρίε και κύριοι, αυτό είναι και επικίνδυνο αυτή η κατασκοπία. Ε, πρέπει λοιπόν να το δούμε πολύ σοβαρά. Και ε, το θέμα των παλαιότερων εκδοχών. Ε, κοιτάξτε, ε, σε όλες τις πολιτικές ομάδες διαπιστώθηκε αυτό που δεν θέλουμε να έχουμε στην άκτα. Και καλέσαμε την Κομισιόν να το εξετάσει το θέμα, να καταλήξει. Τώρα λοιπόν αναφέρεται ότι παλαιότερες εκδοχές όπου περιλαμβανόταν το τι δεν μας αρέσει, αυτές να επανέρχονται. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα όπου η Κομισιόν πρέπει να τοποθετηθεί με σαφήνεια. Δηλαδή να πει με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν είναι δυνατόν να επανέρχονται παλαιότερες εκδοχές για να καταλήξουμε στη σημερινή ερμηνεία. Και κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ, ε, αυτό που είπε ο κύριος Αρίφ, πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τη διαφάνεια και τη συνθήκη της Λασσαβόνας. Και μόλις ετέθη αυτή σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010, όλες οι πολιτικές ομάδες επέκριναν την έλλειψη διαφάνειας. Έκτοτε λοιπόν έχουν γίνει πάρα πολλά. Είχαμε πολλές ε, συζητήσεις ε, και στην Ολομέλεια και το 2010 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Ήταν γνωστή η διαδικασία και έγινε ο εισηγητής ο κύριος Αρίφ. Και με ο συντονιστής παρετήθηκε γιατί ήθελε να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές ε, στην Γαλλία και ο εισηγητής παρετήθηκε. Πάει και αυτός. Και τώρα τι λέμε, θέλουμε την συμφωνία της Άκτα ε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την άκτα. Και αυτό που ως ΕΛΚ επικρίνουμε δρυμύτατα είναι, μισό λεπτό, ότι εδώ και τέσσερις μήνες ε, είχαμε έναν εισηγητή, τον κύριο Ρίφ, και τέσσερις ολόκληρους ε, μήνες το θέμα αυτό δεν παρουσιάστηκε σε καμία μερίσια διάταξη της Επιτροπής μας. Γι' αυτό λοιπόν ως ΕΛΚ επιμείναμε εμείς να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα. Επιτέλους να γίνει μια δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό. Και αυτά του μύθου και του κυρίου Αρίφ, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανηλικρίνη που έζησα ποτέ εδώ στο Κοινοβούλιο τελευταία 8 χρόνια και νομίζω ότι θα βοηθούσε όλες αν μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Πριν θα δώσω το λόγο μάλλον πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Επίτροπο και μετά στον David Μάρτιν. Επιτρέψτε μου όμως επίσης να σας ε, παρουσιάσω και τη δικιά μου τη θέση για διάφορα θέματα αρχής. Πρώτα απ' όλα, βαζόμενοι στη γνώση, στην έρευνα, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ενισχύσουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι η γνώση είναι το πιο, πιο βασική πρώτη για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, η συνεργασία είναι επίσης ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε υψηλή προστασία και καλή εφαρμογή της προστασίας των, ε, της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Όντως υπάρχει και θέμα δικαιωμάτων ε, των δημιουργών των ερευνητών, των συγγραφέων, των μουσικών κτλ. Πρέπει να προστατεύονται. Η παραποίηση και η πειρατεία προϊόντων πρέπει να καταπολεμάται. Έπειτα δεν βλέπω εγώ καμία διαφορά στο να ανοίξουμε ένα μαγαζί στις Βρυξέλλες κάποιος και να πουλάει παραπημένα προϊόντα και να ανοίξει κάτι αντίστοιχο στο διαδίκτυο. Για μένα είναι το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη μία περίπτωση και την άλλη. Τέλος, κατά τη γνώμη μου, μια κακή ερμηνεία της άκτα δεν ε, πλήττει ατομικά δικαιώματα ή ελευθερίες. Κατόπιν αυτό θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Τεγκούχ να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτή τη φορά θα περιορίσω και το δικό σα το χρόνο. Συνήθω δεν το κάνω, αλλά θα το κάνω. Και μετά θα δώσω το λόγο στον συγκεκριτή. Τι, θέλετε ανάποδα να τα κάνω. Καλά, τότε θα δώσω το λόγο πρώτα στον Ντέβιτ Μάρτιν και μετά στον Επίτροπο. Στο στάδιο αυτό δεν θα επανέλθω επί τη ε, ουσία, οπότε αυτά θα τα απαντήσει ο Επίτροπο. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ένα πράγμα και να ζητήσω και την έγκριση της Επιτροπής μας για τη στρατηγική που θα ακολουθήσω. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της συζήτησης, ο Καντήφα πρέπει να φύγει. Αλλά Βλέπετε πριν από λίγες εβδομάδες μας υπευλήθη το θέμα. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε. Θέλω λοιπόν η Επιτροπή μας, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, αλλά να δούμε μήπως έχει κανείς αντίρρηση. Θέλω λοιπόν να συμφωνήσετε να έχουμε ένα ψήφισμα ε, μετά να έχουμε το δικαστήριο, μετά να έχουμε την Ολομέλεια, να δεχτείτε δηλαδή να πρόκειται για μια προσωρινή έκθεση που θα ετοιμάσουμε όσον αφορά την άκτα. Αν συμφωνείτε, θα ξεκινήσω να δουλεύω ακριβώς με αυτά τα δεδομένα. Καλώς. Ευχαριστούμε, τον το Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Και σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε, πότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, λίγα λεπτά. Πρώτα απ' όλα για το θέμα του απορρίτου. Το απόρριτο, γύρω από το οποίο έγιναν και διαπραγματεύσεις. Εγώ είμαι επίτροπος για το εμπόριο από το Φεβάριο του 2010. Και ευθύς εξ αρχής ζήτησα από τις πλευρές που συμμετείχαν στην διαπραγμάτευση να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Δεν ήταν εύκολο. Δημόσια δηλαδή, έτσι. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που ήθιστε να συμβαίνει στις διεθνείς συμφωνίες. Καλός ή κακός, οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν και δεν ενημερώνεται το κοινό για αυτές, δεν γίνονται ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ το ζήτησα και αυτό έγινε. Δεύτερον, μεταφέραμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δώσαμε πολλά καινούρια έγγραφα, τοποθετήσεις, ό,τι είχε ετοιμαστεί εστάλησαν αμέσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φαντάζομαι ότι δεν τα διαβάσατε όλοι όλα, γιατί πρόκειται για κιλά χαρτιού που αν είχαν τυπωθεί βέβαια, εντάξει δεν λέω ότι τυπώθηκαν, που θα έπρεπε να τα διαβάσετε και δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο για να διαβάζει κανείς. Ίσως. Τρίτον, το Κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες μόνο έλαβε το έτοιμά μας. Εξάλλου δεν μπορούμε να σας υποβάλουμε κάτι αν προηγουμένως δεν έχει υπάρξει μετάφραση και δεν είναι έτοιμο όλα. Αλλά τίποτα δεν σας εμπόδισε να το συζητήσετε και πιο πριν. Εκτός ίσως από την γαλλική προεκλογική εκστρατεία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι δικιά μου ευθύνη, ε, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε πιο σωστοί γι' αυτά. Τώρα γιατί ε, ζήτησα τα σχέδια τοποθετήσεων να γίνουν γνωστά είναι γιατί όντως δεν πρόκειται για μια συνήθη εμπορική συμφωνία. Τεχνικά μιλώντας είναι εμπορική συμφωνία, αλλά έχει να κάνει πολύ περισσότερο να κάνει με τις θεμελιώδεις ελευθερίες από ότι οποιαδήποτε άλλη εμπορική συμφωνία. Η άκτα δεν είναι το ίδιο με τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και ήθελα να είμαστε πιο ανοιχτοί. Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι πολλά πράγματα που αναφέρονται μπορεί κανείς να τα δει έτσι γενικά. Ο όρος ας πούμε commercial skill, η εμπορική ιδιότητα. Όντως υπάρχουν ε, πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με νομολογία. Γιατί η ιδέα αυτή του commercial skill που λέει ότι έχει να κάνει με άμεσα ή έμεσα εμπορικά πλεονεκτήματα είναι κάτι που σύχθη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με την οδηγία Lending του 1992. Και μετά επιβεβαιώθηκε και σε άλλη οδηγία το 2006. Χρησιμοποιήθηκε μια νέα ένας νέος ορισμός το 2004 και έπειτα υπάρχει και το άρθρο 61 της συμφωνίας TRIPS, είναι η συμφωνία του ΠΟ έτσι για την πάλι πνευματική ιδιοκτησία. Εκεί το άρθρο 61 λοιπόν λέει ότι τα μέλη θα προβλέψουν κυρώσεις και τα λοιπά να προβλέπονται σε περίπτωση παραποίησης ή πειρατείας, εφόσον αυτή γίνεται για, σε εμπορική κλίμακα. Η Επιτροπή δεν διαπραγματεύτηκε για το θέμα ποινών της άκτα, τα κράτη-μέλη το κάνανε. Οπότε τα κράτη-μέλη τώρα κάθονται και σχολιάζουν και έχουν παρατηρήσεις για το θέμα για το οποίο τα ίδια διαπραγματεύτηκαν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν που διαπραγματεύτηκαν το ποινικό σκέλος, λέει λοιπόν σε εμπορική κλίμακα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λέει το άρθρο 23 σημείο 1. Κάτι το οποίο έχει ετοιμαστεί από την ε, νομολογία πάρα πολύ προσωπικά και δεν μιλάει, αποκλείει δηλαδή τους καταναλωτές που δρούν καλή την πίστη. Όταν ετοιμάζεται μία σύμβαση, μία συμφωνία, υπάρχουν διάφοροι όροι, τους οποίους εξηγείται στην αρχή της συμφωνίας. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με έναν όρο, ο οποίος ορίζεται συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οπότε εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση για την άκτα. Η άκτα έχει να κάνει με την εφαρμογή, με τη θέση σε ισχύ, δεν έχει να κάνει με την νομοθεσία. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα με την νομοθεσία, πονέρθουμε αργότερα σε αυτό μου θέλετε, αλλάξτε το, είσαστε το κοινοβούλιο. Η Επιτροπή, άμα κάνετε τέτοια πρόταση, θα προχωρήσει. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω τροποποίηση στη θεμελιώδη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν μου το ζητήσετε εσείς. Στα χέρια σας είναι λοιπόν αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι α, δεν συμφωνούμε με την νομοθεσία αυτή ενώ υπάρχει το θεμελιώδες δίκαιο που το περιλαμβάνει. Αν θέλετε να το αλλάξετε, αλλάξτε το. Εσείς έχετε δικαίωμα αρνησικυρία σε αυτό. Δεν μπορούμε τίποτα να βάλουμε εκεί αν εσεί δεν συμφωνείτε. Είναι δικιά σα ευθύνη. Αν υπάρχει κάτι που δεν σα αρέσει, είναι δικιά σα ευθύνη. Εσεί το έχετε ψηφίσει αυτό. Οπότε να βάλουμε τι ευθύνε εκεί που είναι. Τώρα για τα γνώσιμα φάρμακα. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά προβλήματα. Από τη μια μεριά υπάρχει η Συμφωνία Άκτα και από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι συζητήσεις που γίνονται στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και μερικέ φορές υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο. Υπήρξαν κατά το παρελθόν προβλήματα πάλι από τα κράτη-μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί γιατί στις κάτω χώρε έγινε μια κατάσχεση γεννόσιμων φαρμάκων και μια φορά και στη Γαλλία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί πια, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει τις οδηγίες σε σχέση με τους τελωνιακούς ελέγχους. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν πια έλεγχοι σε σχέση με τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Αλλά το θέμα είναι η παραποίηση και η πειρατεία. Και εγώ παίρνω εκατοντάδες email για τα φάρμακα το γεγονός ότι δεν θα γίνεται πια ο έλεγχος παραπημένων φαρμάκων, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στον υπονάπτυξη κόσμο. Πάνω από 10% των γενώσιμων φαρμάκων είναι παραπημένα. Μπορεί να υπάρχουν φάρμακα για το AIDS για παράδειγμα, αλλά τελικά είναι απλώς πλασεμπό, δεν είναι τίποτα δηλαδή. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί νομίζουν ότι παίρνουν φάρμακα που τους προστατεύουν για παράδειγμα από την εξέλιξη της ασθένειας του AIDS ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπότε γιατί εμείς, χωρισμένοι μέλη δηλαδή, να μην κάνουμε ελέγχους σε ό,τι φτάνει στα λιμάνια μας, στα σύνορά μας, για να δούμε μήπως είναι επικίνδυνο για την υγεία. Δεν θα έπρεπε. Ειλικρινά θέλω μια σοβαρή απάντηση γι' αυτό και από το Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τώρα. Τι θα κάνει, τι θα ελέγξει, τι γνωμοδότηση θα μας δώσει. Εννοείται, εκείνοι θα το αποφασίσουν εμείς, ερωτήσεις τους κάνουμε και θέλουμε να μας απαντήσουν. Κύριε Ζαντό, πήραμε την απόφαση να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά αυτό δεν αποτελεί ε, κομμάτι της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας. Όχι, είναι κομμάτι που αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό το κάναμε τώρα. Έπειτα, ο πρόεδρος της Επιτροπής σας το ήξερε και ο εισηγητής. Ε, πήρα τηλέφωνο τον Ντέιβιντ και του είπα, κοίταξε, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά αν εγώ θέλω να το κάνω ω επίτροπο, πρέπει να το περάσω από το Σώμα των Επιτρόπων. Δεν μπορώ να το κάνω από μόνο μου. Πήγα λοιπόν στο Σώμα των Επιτρόπων και ακούστηκε ότι πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι απόφαση του Σώματο των Επιτρόπων. Χάσατε τίποτα εξάλλου επειδή δεν το ξέρατε από πριν. Και εσεί είχατε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έτσι. <clears throat> το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να δεχτεί αιτήματα και από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή και από το Σεβούλιο και από οποιαδήποτε χώρα μέλος. Οπότε δεν βλέπω γιατί διαμαρτύρεστε. Τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τι θα κάνει. Ε, φυσικά αναφέρεται στη συνθήκη και μέρος της συνθήκης είναι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό που επανελειμμένα κατά το παρελθόν έχει κάνει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ότι ελέγχει κατά πόσο το παράγω δίκαιο συνάδει με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για παράδειγμα με το δίκτυο ΣΑΒΑ κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα κοιτάξει μόνο τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτά καθ' αυτά, αλλά θα μπει στο βάθος της υπόθεσης και θα δει τι μπορεί να συμβεί με το παράγω δίκαιο. Εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφανθεί ουσιαστικά, δεν θα πει απλώς ε, είναι ή δεν είναι σύμφωνο, Διαβάστε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ σπάνια βρήκα μία που να είναι λιγότερο από 25 σελίδες. Συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερες. Οπότε θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνονται και την συμφωνία αυτή. έχει να κάνει επίση και με το δικαίωμα ιδιοκτησία. έτσι γιατί και η πνευματική ιδιοκτησία είναι ιδιοκτησία. Σίγουρα θα αναπτύξουν πολύ περισσότερο την ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών. Και εκτός από την άκτα είναι γενικότερα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε αυτή την απόφαση. Το επιχείρημα τώρα που επίσης ήρθε σε πολλές περιπτώσεις είναι «Μα δεν συζητάτε με τους σωστούς εταίρους». Δεν είναι για την παραποίηση. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς θα σταματήσουμε την παραποίηση και την πειρατεία. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε και με τις αναδυόμενες οικονομίες. Αλλά βλέπετε, δεν το θέλουν. Γιατί αυτοί που πραγματικά θέλουν να προστατευτούν τα δικαιώματα διοκτησία είναι οι πιο όριμε οικονομίε. Οι αναδυόμενε προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν όσο μπορούν την πνευματική διοκτησία χωρί να πληρώσουν. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε αυτό με την Κίνα. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν και με άλλε αναδυόμενε οικονομίες, οι οποίε τώρα πια, ε, ευκαιρία σας το λέω, είναι όριμε οικονομίες. Άρα λοιπόν δεν έχετε συνομιλητή από τις αναδυόμενες ε, οικονομίες, μπορείτε όμως να σταματήσετε τα παραπημένα προϊόντα στα σύνορα. Και όταν έχουν και εκείνες οι χώρες όριμη οικονομία, μπορούμε να συζητήσουμε και μαζί τους παρετέρω. Έπειτα, για το θέμα του ουσιαστικού δικαίου. Έχω να πω ε, κάποια πράγματα, θα τα πούμε σήμερα το απόγευμα. Χρειάζεται σίγουρα ενημέρωση. Η Επιτροπή φυσικά και μπορεί να έρθει με κάποιες προτάσεις. Έχετε και την οδηγία για την ε, θέση σε ισχύ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο τώρα το έχουμε μια δεκαετία. Ίσως θα πρέπει να αλλάξει κάτι, να υπάρξει ενημέρωση. Αλλά εσείς ως κοινοβούλιο πρέπει και εσείς να αναρωτηθείτε μήπως υπάρχει πρόβλημα με τις εθνικές νομοθεσίες και για τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί σε όλα τα μέλη που παίρνω ε, πάντα μου λένε αυτό, ότι τρία λάθη και μετά ποινή. Αυτή η ιστορία του three strike είναι κάτι που υπάρχει στη Γαλλία στην νομοθεσία. Και πρέπει και εσείς να αναρωτηθείτε λοιπόν για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή είναι μια νομοθεσία η οποία έχει αποφασιστεί προκειμένου να πάλι σε εφαρμογή ευρωπαϊκές οδηγίες. Άρα και εσείς κάτι μπορείτε να κάνετε εδώ. Στη συμφωνία ΑΚΤΑ λέει ότι δεν μπορείτε να έχετε τα three strike. Δεν μπορείτε αυτό σε διεθνέ επίπεδο να το χρησιμοποιήσετε. Ναι, αλλά σε εθνικό επίπεδο επιβάλλεται. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ μεγάλων χωρών όπως η Γαλλία. Να το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Μια τελευταία παρατήρηση τώρα, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει και εγώ να τηρήσω το χρόνο που μου δώσατε. Λέτε ότι μας έρχεται πολύ αργά και ότι υπάρχει ήδη συμφωνία. Ότι πρώτα θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το έμπρακτο και μετά να έρθουμε εδώ. Τώρα, αυτή είναι μια πολύ περίεργη παρατήρηση. Γιατί το Συμβούλιο εξέτασε τη συμφωνία και συμφώνησαν ομόφωνα, αλλά όχι μόνο το Συμβούλιο ως θεσμός, αλλά και τα κράτη-μέλη ομόφωνα συμφώνησαν γιατί πρόκειται εδώ για μια μεικτή συμφωνία που πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα ποινικά κεφάλαια. Άρα υπάρχει ομοφωνία. Και ξαφνικά αρχίζουν και το ξανασκέφτονται. Τι σημαίνει, δεν κάνανε καλά τη δουλειά του ε, στην αρχή. Τι σημαίνει, ότι τώρα ξύπνησαν. Τώρα κατάλαβαν ότι υπάρχει κάτι που τους ενοχλεί. Μα δεν είναι σοβαρός τρόπος δουλειάς αυτός. Και όλη η ιδέα που λέει να ξαναρχίσουμε τη δουλειά μας, εντάξει μπορεί, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να ξαναρχίσουν τη δουλειά τους από την αρχή και όχι εμείς. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται έτσι η ανταλλαγή απόψεων. Θα έχουμε και δεύτερη ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα το απόγευμα στο εργαστήρι που είναι ανοιχτό για όλους. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγκούχ που ήρθατε και και σήμερα. Τώρα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Ποια σημεία θα παραλείψουμε, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Και θα τα αφήσουμε δηλαδή για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, προσωπικά κρίνω ότι οφείλουμε να αποδώσουμε προτεραιότητα στο σημείο 21, 22, 24, Θα αρχίσουμε με το θέμα του Ρόμπερτ Στέρντι που είναι εισηγητή. It's Πρόκειται για κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλιβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος γιατί μας πιέζει, σας παρακαλώ, πρόεδρε, διακόπτη ο μιλητή. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα σημεία αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση, δηλαδή το 25 και 26. What, is that we... Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουμε. Ας δούμε ποια μπορούμε να ολοκληρώσουμε και τα υπόλοιπα θα εγγραφούν στο, στην μέση διάταξη επόμενη συνεδρίαση. Σημείο 22. Δεν είναι εδώ ο Ρόμπερτ Στέρντι, αλλά μου είπε ότι θα αντικατασταθεί από τον κύριο Κάμπελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ, ε, μπορείτε να, προσέξτε τι λέει ο αντικαταστάτης του εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Στέρτη μου έδωσε τις ε, σημειώσεις του για να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για αυτό το θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω μια συμφωνία που ήταν σε ισχύ το χρονολογείται από το 2007 για εμπόριο ορισμένων ειδών χάλιβα χρειάστηκε να ε, καταργηθεί διότι εισήλθε στον ΠΟΕ η Ρωσική Ομοσπονδία. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο Ρόμπερτ Στέρντ είναι το εξή. Ε, πιστεύει ακράδαντα ότι ο ΠΟΕ είναι και ο καλύτερο ε, εγγυητή θεματοφύλακα ε, των κανόνων ενό πολυμερού εμπορικού συστήματο. Έθεσε την εξή ερώτηση στον Πασκάλ Λαμή σχετικά με την εποπτεία τη προσχώρηση τη Ρωσική Ομοσπονδία στον ΠΟΕ και αν υπήρξε συμμόρφωση με του κανόνε και αν υπάρχει ακόμη συμμόρφωση με του κανόνε. Ε, και έλαβε την, ε, εξέφρασε την ανησυχία ότι δεν θα τηρήσει η Ρωσία τους ε, κανόνες και προτείνει στον κύριο Λαμία ετησίω να υποβάλλεται έκθεση παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το αν σέβεται και τηρεί τους κανόνες η Ρωσική Ομοσπονδία ή όχι. Δεν θέλησε να δώσει ούτε υπόσχεση να αναλάβει δέσμευση ο Επίτροπος. Πάντως ο Ρόμπερ Στέρντι πιστεύει ότι αυτή η τετραετής περίοδος πιστευει οτι αυτη η τετραετη σε περιοδος οπως και για την Κίνα παρά μακρά για την Ρωσία και επιμένει ετησίω να υποβάλλεται η έκθεση και όχι κάθε τέσσερα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης το έχετε στους ε, φακέλους σας και τώρα θα ακούσουμε τους ε, σκιώδεις. Ε, Δεβάντερε, από το ΕΛΚ δεν θέλετε. Ποιος θέλει το λόγο. Θέλετε να αρχίσει Σιλβάνα Κόχμερη από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κάμπο, ευχαριστούμε που αντικαταστήσατε τον κύριο Στέρτη και μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εγώ συμφωνώ με το σχέδιο αυτό αυτό είναι ένα επίσημο αίτημα ουσιαστικά για το οποίο πρέπει να τοποθετηθούμε. Εγώ προσωπικά θα είχα όμως και κάποιες ανησυχίες ως προς το επεξηγηματικό σημείωμα που δια, ε, μας διαβιβάζεται. Ο Ρόμπερ Στέντι ζητάει ετήσια έκθεση από τον ΠΟΕ και πιστεύω ότι αυτή η διατύπωση πρέπει να είναι ρητή μέσα στο κείμενο. Όχι μόνο ότι επιθυμούμε να υποβάλλεται αιτήσια η έκθεση, αλλά και ότι επιθυμούμε να διεξαχθεί η διεξοδική ανάλυση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σημαίνει δηλαδή για τη χαλιβουργική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το να εγκαταλειφθεί αυτό το σύστημα των ποσοστώσεων. Εγώ πιστεύω ότι είναι θετικό, αλλά με υπέρ της απελευθέρωσης, αλλά καλό είναι να ξέρουμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Οπότε μελέτη αντικτύπου για την ε, ε, βιομηχανία χαλιβουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς ε, θα επηρεαστεί και αν χρειαζόμαστε κάποιο είδου μεταβατική περίοδο ή κάποιους ειδικούς μηχανισμούς διασφάλισης, όπως ισχύει σε άλλου τομεί και με άλλε χώρε. Έκανε κάποιε εκτιμήσει αρχικέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το όφελο που θα αποκόμιζε η χαλιβουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κατάργηση. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν κατάλαβα, δεν είναι σαφή η απάντηση στα μάτια μου. Οπότε καλό θα ήταν μέσα στο επεξηγηματικό και διαβαστικό σημείωμα να συμπεριλάβουμε ρητά αυτή τη μνήμα ότι ζητάμε δηλαδή ε, υποβολή αιτήσια έκθεση και μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή ναι. Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Τώρα, σοσιαλιστές. Σιγητής, και ο από πλευρά των ε, σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Με την ιδιότητα του σκιώδους ε, εισηγητή, Μπορώ να τοποθετηθώ και να σας πω ότι θα εγκρίνουμε αυτή την έκθεση. Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει προσχωρήσει στον ΠΟΕ και άρα είναι ε, άχρηστο ε, πλέον ο κανονισμός. Το να διατηρηθεί δεν ισχύει, παραβιάζει και τους κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, πιστεύω και θα ήθελα ε, ο, ο ΠΟΕ να παραμείνει, να εξακολουθήσει να είναι ο βέλτιστος δυνατός εγγύητης και θεματοφύλακας των ε, κανόνων του πολυμερούς εμπορίου. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μία διόρθωση θα κάνω. Πάτε Ζαλεύσκη, είναι ο Σκιώδης από το ΕΛΚ. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας έδωσα πρώτος. Το... ο μιλητής μιλάει εκτός μικροφόρων, δυστυχώς δεν τον ακούμε. Uh, uh, um, Ευχαριστώ. Πολύ θετικό που η Ρωσία επιτέλους ε, προσχωρεί στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όμως ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει υπερβολική πλεονάζουσα ρωσική ικανότητα στον τομέα του χάλιβα από πλευρά Ρωσία πάνω από 40 εκατομμύρια τόνου. Καταλαβαίνετε πως κατακλείζεται η αγορά. Ε, δεν γίνεται να μην προβλέψουμε προστασία, καταφύγιο για την ευρωπαϊκή χαλιβουργία. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ε, μετά την κατάργηση των ποσοστών να εκτιμηθεί η, ε, επακριβώς η κατάσταση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει στην αγορά και ακόμη πιο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί την άρση υπολοιπόμενων φραγμών και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ε, παραδείγματος χάρη για ε, τις αγορές πρώτων υλών. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε διεξοδική ανάλυση της αγοράς ε, για τις ε, πρώτες ύλες, για την ε, χαλιβουργία, για την δημόσια παρέμβαση στην αγορά και τα μέτρα προστατευτισμού καθώς και το καθεστώς και το γενικότερο περιβάλλον για τις άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις στη Ρωσία για να έχουμε μια σφαιρική εντύπωση της κατάστασης. Ευχαριστώ τώρα από πλευρά των Πρεσίνων, Πρόεδρε. Αναγνωρίζουμε ότι ε, συντρέχει νομική υποχρέωση να καταργήσουμε αυτόν τον κανονισμό σχετικά με τις, ε, τους περιορισμούς στο εμπόριο. Ε, θέλαμε όμως να τονίσουμε ότι στους παραγωγούς χάλιβα και η Ρωσία ούτως ή άλλως είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι από όλους τους παραγωγείς ε, ανά τον κόσμο ε, η ρωσική χαλιβουργία είναι η πλέον ρηπογόνα ως προς τους, τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Η παραγωγή ενδέχεται να αυξηθεί έτσι περαιτέρω και μας ανησυχεί αυτό για την συνέχιση της διαδικασίας, δηλαδή η εμπορική πολιτική ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα αντιβαίνει στην περιβαλλοντική και άλλες πολιτικές της, της Ένωσης και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί αυτό το θέμα στην υποδιαπραγμάτευση εταιρική σχέση και την υποδιαπραγμάτευση νέα εμπορική συμφωνία με τη Ρωσία. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή? Who will speak on behalf of the Commission? Yes, the floor is yours. For the sake, for the record, could you identify? Μπορείτε να μας συστηθείτε για τα πρακτικά. Ναι, Πρόεδρε. Πέτρος Ερμένης από τη Γενική Διεύθυνση Trade. Ευχαριστώ τους ε, ομιλητές ε, για τα σχόλιά τους. Όπως αναγνώρισαν όλοι, η κατάργηση του κανονισμού για τις ποσοστώσεις για, κάποια, ε, για την εισαγωγή χαλιβουργικών ειδών από την Ρωσική Ομοσπονδία είναι λογική απόρρια της προσχώρησης της χώρας των ΠΟΕ. Ε, φυσικά, η κατάργηση θα λάβει χώρα όταν η Ρωσία αναλάβει τη θέση του πλήρους μέλους του ΠΟΕ, αναμένουμε δηλαδή το καλοκαίρι να γίνει αυτό. Μέχρι τότε θα συνεχίσουν ε, να εφαρμόζονται οι ποσοστώσεις και η διαχείρισή τους ε, θα διέπεται από τον ε, τωρινό κανονισμό. Σε σχέση τώρα με την κατάργηση του κανονισμού, είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΠΟΕ, ακόμη και για την, τον τομέα παραγωγής χάλιβα, για τη χαλιβουργία δηλαδή, και ε, την ε, μείωση των δασμών ε, για τελειοποιημένα χαλιβουργικά προϊόντα και όπως ανέφεραν και κάποιοι ομιλητές στις πρώτες ύλες θα μειωθούν οι εξαγωγικοί δασμοί ταυτόχρονα που εφαρμόζει η Ρωσία για την εξαγωγή παλιοσίδερων. Επίσης θα, το καθεστώς θα ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες του ΠΟΕ Και φυσικά χρειαζόμαστε, ε, χρειάζεται να εγγράψουμε αυτή την κατάργηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ακούσαμε τους, ε, τις παρεμβάσεις, ε, ακούσαμε την ερώτηση αν θα αυξηθούν με την κατάργηση του κανονισμού οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Έχουμε ήδη συζητήσει με την Επιτροπή Ίντα αυτό το θέμα πριν από λίγους μήνες είναι προφανές ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τις εξελίξεις και θα είναι διπλή αυτή η παρακολούθηση. Πρώτον, θα ενεργοποιήσουμε αυτή την ε, ομάδα επαφής για το Χάλιβα, έτσι ονομάζεται, όπου θα συσκεφτούν δηλαδή εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθώς και εκπροσώπους του κλάδου ε, αμφωτέρων ε, των πλευρών η πρώτη συνεδρίαση θα λάβει χώρα σε λίγους μήνες αυτής της ομάδας επαφής για να παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση και συλλέγουμε ταυτόχρονα διάφορα στατιστικά στοιχεία. Θα συνεχιστεί η συλλογή των στοιχείων για να παρακολουθούμε την ε, κατάσταση. Αυτά που μας δείχνουν οι στατιστικές μέχρι στιγμής και αυτά που μας έδειξαν πέρυσι ήδη και συνεχίζουν να δείχνουν φέτος είναι ότι η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί πλήρως ε, τις ε, ποσοστώσεις που έχει δυνάμει της ε, διμερούς συμφωνίας. Το 2010, για να έχετε μία ιδέα, η Ρωσία χρησιμοποίησε 61% της συνολικής ποσόστοσης για προϊόντα χάλιβα που έχει στη διάθεσή της αληθεύει ότι κάποια προϊόντα για τα οποία το ποσοστό απορρόφησης είναι υψηλότερο, κυρίως για τις θερμές χαλίδινες ράβδους, ε, ε, ε, είναι χαμηλό, αλλά μπορούμε να φτάσουμε και σε ποσοστό 93%. Το 2011 το ποσοστό ήταν 55% για γενική χρήση και 77% χρήση στα πιο σε εισαγωγικά ευαίσθητα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη τα θερμά ελάσματα. Και συντρέχει ο κίνδυνο μετά την καταργήση του κανονισμού να αυξηθούν οι εξαγωγέ τη Ρωσική Ομοσπονδία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ το παρόν όμω τα στοιχεία δεν μα επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε μια τέτοια τάση. Ως προς το θέμα του αν η Ρωσική Ομοσπονδία θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της βάση νομοθεσία του ΠΟΕ, ε, πρόεδρε, ε, θα αναφέρω τα εξής. Η, η έκθεση που υποβάλαμε για τις ε, επενδύσεις και για το εμπόριο για το 2012 που κατατέθηκε σήμερα ε, ενώπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και φυσικά διαβάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα κεφάλαιο σχετικά με την ε, προσχώρηση της Ρωσίας. Μίλησε, μιλάμε για άρση κάποιων φραγμών από πλευράς Ρωσίας για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και φυσικά παρακολουθούμε στενά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ρωσία και η ομάδα επαφή ε, για αυτά τα προϊόντα. Του όλου θα ενημερώσει κατά το ΔΕΜ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που ελέγχθησαν και συμφωνώ με αυτό που ελέγχθη σχετικά με τη συμφωνία του ΠΟΕ γιατί ε, αυτό έχει σχέση και με αυτό που πιστεύει ο κύριος Στάοντι. Νομίζω θα υπάρξει μια συζήτηση στην Ολομέλεια από αυτού και εκεί θα ληφθούν υπόψη πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Θέλω να πω ότι όσον αφορά τους κανόνες του Κοινοβουλίου δεν, με βάση αυτούς δεν μπορούμε να αλλάξουμε το επεξηγηματικό σημείωμα για να λάβουμε υπόψη μας αυτά που ελέγχθησαν. Πάντως ε, θα γίνει αυτή η συζήτηση και θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις. Αυτό μου είπαν. Θα ληφθούν υπόψη, υπόψη παρατηρήσεις, αν όχι εδώ, σε κάποιο άλλο σημείο. Επόμενο βήμα ε, στη διαδικασία είναι η διορία για την κατάθεση τροπολογιών αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Μην το ξεχνάτε αυτό, γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό το να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πάμε στο 21 που και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να αποφασίσουμε γι' αυτό σήμερα γιατί αφορά τις ε, τροπολογίες ε, στην αποκαλούμενη συμφωνία Omnibus του και αφορά στην προσαρμογή του ε, νομοθετικού κεκτημένου της ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, προς την διαδικασία των κατεξουδότηση πράξεων και τις εφαρμοστικές διατάξεις με βάση τη διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας. Οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Ο αριθμός των τροπολογιών δεν είναι τόσο μεγάλος, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση αυτού του κανονισμού. Αρμόδιος εισηγητής είναι ο κ. Γκλασίτ από τους σοσιαλιστές θα αντικατασταθεί από τον κύριο Μπέρντ Λάγκα από την ίδια πολιτική ομάδα. Μπέρντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τώρα κατά πόσο μπορώ να τον αντικαταστήσω δεν το ξέρω αλλά ε, θα προσπαθήσω να σας ανακοινώσω τις σκέψεις του. Καταρχήν, ο Γιούρν Λάχτφριντ θέλει να ευχαριστήσει όλους ε, για την ε, καλή συνεργασία, κυρίως την τώρα, κυρία Ρόβολτ, γιατί εντωμεταξύ συμφώνησαν σε όλα σχεδόν τα σημεία και ως εκ τούτου προκύπτει ευρεία συνένεση. Υπάρχουν βέβαια πολλά τεχνικής φύσεως θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι σημαντικά αυτά, γιατί αφορούν ε, στην διάδοχο, στον διάδοχο κανονισμό του κανονισμού περί επιτροπολογίες και εδώ εξετάζονται κυρίως η κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, αυτές ε, είναι καθοριστική σημασία για την δυνατότητα της συναπόφασης του Κοινοβουλίου. Τώρα, παρατηρήσει επί της ουσίας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι αποσύρουμε το δίκαιο Μάλλον ότι με τις κατεξιδότητες πράξεις μπορούμε να αποσύρουμε κάποιες ε, νομοθετικές διατάξεις. Ε, οι διορίες ε, αναβάλλονται από δύο σε τέσσερις μήνες και ο κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά και αυτός παίρνει το ίδιο, την ίδια παράταση. Αυτό που νομίζω είναι καθοριστική σημασία είναι το εξής ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να συμπεριληφθούν στις διαβουλεύσεις κατόπιν τούτου μπορούμε να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Μικρές διαφορές υπάρχουν στο ερώτημα πώς ακριβώς ορίζονται οι εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου ε, και ο κύριος Λάιχτφριτ επιθυμεί να προβάλλει εμφατικά ε, το ότι αυτοί ε, να μπορούν να καλούνται και αυτόνομα για να υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία ακριβώς ε, όπως γίνεται και με τους εμπειρογνώμονες της αγοράς. Για τα θέματα αυτά θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η επόμενη συνάντηση των σκιωδών συντονιστών είναι την Τρίτη στο Στρασβούργο σε 6 ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστούμε, ε, Μπέρντ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια από αυτού, από άλλα μέλη της Επιτροπής. Ας πάμε τώρα ε, στην Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας εκ μέρους της Επιτροπής τον εισηγητή, ε, το σκιώδη εισηγητή και όλους τους ε, συναδέλφους ε, που δούλεψαν για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ για την πρόοδο που επιτεύχθηκε. Εμείς έχουμε που θα τα κάνω πολύ σύντομα και αφορούν στο σχέδιο της έκθεσης και στις περαιτέρω προτινόμενες τροπολογίες. Δεν θα επαναλάβω βέβαια όλα τα σχόλια ε, τα οποία έγιναν ήδη στην τελευταία επιτροπή. Τα πρώτα σχόλια αφορούν στην ε, νομοθετική τεχνική που προτείνεται. Ε, ο εισηγητής προτείνει να συμπεριλάβουμε εδάφια και ο Σκιώδης Συγητής λέει ότι θα πρέπει να αρθούν όλες οι αναφορές στο σύστημα επιτροπολογίας του 1999. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη για την κωδικοποίηση αυτών των πράξεων μόλις έχει ολοκληρωθεί η Omnibus 1 και η Omnibus 2. Βέβαια, ε, για λόγους συνέπειας με την Omnibus 1, αυτό θα γίνει στην Omnibus 2 και αυτό θα στηθεί περιττέρω στην τριμερή συνάντηση. Το δεύτερο θέμα που θέλουμε να σας επισημάνουμε είναι το θέμα της ε, κατά πόσον πρέπει να υπάρχουν δύο επιπρόσθετες προτάσεις για, τα, για τις πράξεις σχετικά με τους εμπειρογνώμονες. Η Κομισιόν προτείνει ότι δεν είναι σκόπιμο να υπάρξει ένας ειδικός κανόνας στον τομέα της εμπορικής πολιτικής ή γενικά να υπάρξει οποιοδήποτε ειδικό ε, κανόνας. Ε, το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά την προετοιμασία της ε, κοινή συμφωνίας και επίσης και στη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν η συμφωνία πλαίσιο και η κοινή συμφωνία είναι ο κατάλληλος χώρος για να συζητηθούν αυτά τα δύο θέματα. Κατόπιν τούτου εμείς προτιμούμε την προσέγγιση ε, της εσκιώδου συγγήτριας ε, στις ε, τροπολογίες της για όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε ένα τρίτο σύντομο σχόλιο για την τροπολογία υπαριθμών 54, όπου η σκιώδης συγγήτρια προτείνει να μην ε, συμπεριληφθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία κατεπίγοντος για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Η Κομισιόν όμως πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο γιατί έχει σχέση με την κρίση στον τομέα της υγείας και τα φάρμακα. Είναι ε, σημαντικό να διατηρηθεί η διαδικασία κατεπίγοντος. Και το τέταρτο σχόλιο μου αφορά επιπρόσθετες τροπολογίες από το σκιώδη ηγητή για την ε, κατάθεση εισηγήσεων. Ε, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει πίεση στους πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υποπτεύομαι ότι αυτό είναι επίσης σημαντικό για την τριμερή συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, Μπέρντ, δεν έχει να κάνει σχόλιο Μπέρντ. Κατόπιν τούτου μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία η οποία και θα λάβει χώρα ε, στην επόμενη τακτική συνάντησή μας που είναι στις 26 και 27 Μαρτίου. Και εκεί θα ληφθούν υπόψη όλα τα θέματα που έφυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ, που σημαίνει τρία από τα θέματα της σημερινής αντιάταξης από τα 24 που είχαμε να εξετάσουμε στην ημερήσια διάταξή μας, αυτά τα τρία δυστυχώς πρέπει να αναβληθούν για την επόμενη συνάντηση. Ζητώ συγγνώμη από τα μέλη της Επιτροπής, από τους εισηγητές και βεβαίως και από τα μέλη της Επιτροπής που ήρθαν εδώ περιμένοντας ε, να παρέμβουν ε, σε αυτά τα θέματα που, όπως σας είπα, αναβάλλονται. Αλλά τι να κάνουμε, η συμφωνία Άκτα ήταν ε, πολύ σημαντική για μας και έτσι μας έφαγε το χρόνο. Πρόεδρε, είμαι ένας από τους εισηγητές ε, για την αναβολή. Να γίνει η αναβολή στις 26 Μαρτίου, την πρώτη μέρα της επόμενης συνάντησής μας. Εντάξει, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Τελειώσαμε λοιπόν, λέει ο πρόεδρο, τελείωσε η συνάντησή μας. Θα συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα με το workshop, ε, την ομάδα εργασία, που έχει οργανώσει το Κοινοβούλιο για μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.